Λοιπόν, συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη συνεδρίασή μας. Όλοι εδώ είναι νομίζω. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Στην ημερήσια διάταξη να σας πω πως κατόπιν συμφωνίας με τους συγητέ, έγινε μια αλλαγή. Το 20 και το 21 αλλάζουν θέση. Την Τετάρτη δηλαδή, έτσι, την Τετάρτη. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, το αποφασίζουμε. Αλλιώς δεν υπάρχει κάποια επιθυμία αλλαγή της ημερήσια διάταξης. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω να προσπαθήσετε στις παρεμβάσεις σας να λάβετε υπόψη το ε, τη ημερήσια διάταξη. Το γοργόν και χάρη να έχει δηλαδή. Οπότε περνάμε στην έκθεση της κυρίας Γιόρνταν Σίσελη για ε, τα απόβλητα και θα της δώσω τον λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίλη, ε, Ξέρετε πως κάνω λοιπόν, αυτή την έκθεση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα κάνω κάποιες γενικέ παρατηρήσεις και μετά θα περάσω στις τροπολογίες. Συζητήσαμε με τους κοιοδησηγητές τη βδομάδα που μας πέρασε και τέθησαν δύο ερωτήματα. Ένα ε, ουσιαστικό, πώς το, θα μπορούσαμε να, να αναβάλουμε αυτή την έκθεση για κάποια στιγμή αργότερα λόγω του σεισμού στην Ιαπωνία. Οπότε τα ξαναείδα εγώ όλα αυτά και δεν βλέπω να υπάρχει λόγος για να αναβληθεί αυτή η έκθεση. Δεν το βλέπω γιατί θεωρώ πως ε, τώρα θα πρέπει να αντιδράσουμε για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά ε, απόβλητα. Ξέρετε ε, πως ε, το άλλο θέμα γενικής φύσεως αφορά την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, διαδικασία και το πώς θα ληφθούν υπόψη οι δικές μας απόψεις και Ήδη μόλις ε, η βοηθός μου εδώ με ενημέρωσε πως η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελήφθη. Ο κύριος Λάσλο Κιόμπλιγκερ, αναπληρωτής, γενικός διευθυντής ε, της Ουγγρικής Ρυθμιστικής Αρχής είναι επίσης παρόν, είναι ο αρμόδιος στο Συμβούλιο για αυτή την οδηγία και χαίρομαι που είναι εδώ πέρα μαζί μας και έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί του και βεβαίως πρέπει να συνεργαζόμαστε καλά και με το Συμβούλιο. Λοιπόν, για τις τροπολογίες τώρα προσπάθησα να ενισχύσω τις, ε, να ενισχύσω με τις τροπολογίες την πρόταση αυτή θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτές. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία αρχή η οποία εισάγεται και αφορά την ε, ανάκτηση των αποβλήτων και ε, έτσι αντιμετωπίζουμε την ανησυχία του πληθυσμού ο οποίος επιθυμεί ένα σωστό ε, έλεγχο και βεβαίω το δεύτερο θέμα αφορά τα δημοσιονομικά μέσα γιατί θα πρέπει να έχουμε ισχυρότερες οικονομικές απαιτήσει. θα πρέπει να έχουμε βεβαίως και την αρχή του ρηπαίνοντος εδώ πέρα, να έχουμε ισχυρότερο έλεγχο, να υποβάλλονται εκθέσεις ε, στην Κομισιόν και τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα θα πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητα από τις αγορές και τις πολιτικές επιλογές. Γι' αυτό ζητάμε και τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων για να ασκούν κάποια εποπτεία. Η πρόταση λοιπόν της ε, Κομισιόν είναι πάρα πολύ καλή. Θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε το ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν οι περιφερειακές πρωτοβουλίες μια δικαιολογία για να μην υπάρξει ε, η κατάλληλη δράση. Δηλαδή η διάθεση ραδιενεργών υλικών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ως ένα βαθμό να επιτρέπεται. Εδώ υπάρχει ήδη μια οδηγία περί μεταφορών ραδιενεργών αποβλήτων. Στην ε, δε συνάντηση με τους ε, σκιώδες ηγητές διαπιστώσαμε πως ε, μιλάμε πάρα πολύ για τις εξαγωγές αλλά όχι για τις εισαγωγές ραδιενεργού υλικού Και λύσαμε νομίζω αυτό το ζήτημα. Κατόπιν υπάρχουν κάποιες άλλες αποτίσεις όσον αφορά την διαφάνεια. Η διαφάνεια θα πρέπει να υπάρχει και όσον αφορά το ποιος είναι ο κάτοχος της αδείας. Δεν είναι μόνο θέμα ε, νομοθεσίας και ο κάτοχος αδείας πρέπει να υπόκειται σε διατάξεις σε διαφάνειας καθώς η κοινή γνώμη ε, έχει δικαίωμα να λάβει τις ε, πληροφορίες που θέλει αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει να ακούσουμε και τους ειδικού μετά. Μελέτες ασφαλείας αυτά μέχρι στιγμής βέβαια τα παίρναμε πάρα πολύ σοβαρά αλλά άλλαξε και ο κανονισμός στους ορισμούς και στα άρθρα. Οπότε δεν διαγράφηκε το σημείο αυτό, απλά πήγε σε άλλα σημεία. Κατόπιν... Ε, έχει εισαχθεί η αρχή των ελάχιστων δυνατών πυρηνικών αποβλήτων ήδη από την φάση της ε, παραγωγής κατόπιν όσον αφορά τους εργαζόμενους δεν φτάνει μόνο η εκπαίδευση, το να έχουν ε, δεξιότητες ε, κτλ. Χρειαζόμαστε και προσωπικό στον τομέα της έρευνας ε, και της ανάπτυξης. Ο δε κάτοχος της αδείας θα πρέπει να υποβάλει εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και στις αρχές και στα εθνικά προγράμματα θα πρέπει να υπάρξει ένα σαφές σύστημα κατάταξης ραδιενεργών αποβλήτων. Οπότε θα ήθελα να προσθέσω κάποιες ε, τροπολογίες, να πω παραδείγματος χάρη που θέλουμε έναν ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ των ε, σημείων που αφορούν την πυρηνική ασφάλεια και ε, τον, ε, λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, κενά εδώ πέρα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να επικαιροποιούν τα προγραμματά τους με τις εμπειρίες των άλλων κρατών μελών και διεθνών οργανισμών και βεβαίω εδώ υπάρχει και η απέτηση στα εθνικά προγράμματα της ε, ευθύνης ε, η οποία θα πρέπει να καθοριστεί όσον αφορά τα πρόσωπα και τους φορείς. Λοιπόν, για τις τροπολογίες ε, υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης μέχρι αύριο στις 12 η ώρα. Έχετε την έκθεσή μου μαζί με τις άλλες πληροφορίες. Τροπολογίες όπως σας είπα μέχρι αύριο, οπότε είχαμε ήδη πάρα πολύ χρόνο για να προετοιμάσουμε τις τροπολογίες πάνω από τρεις εβδομάδες και με τους ε, σκιώδεις συζητητές θέλουμε να επιτύχουμε όσο δυνατόν περισσότερες συμβαστικές. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να δώσω λόγο στην κυρία Ρόλ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που μας προτείνει στις τροπολογίες της και χαίρομαι για αυτά που δηλώνει σχετικά με τη διαφάνεια και την ανάγκη της εμπλοκής ε, του δημόσιου τομέα ε, και της αρχής του ρηπαίνων πληρώνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, καλό είναι να μην αφήσουμε παραθυράκια και συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ καλό που αναφερόμαστε και στα στρατιωτικά απόβλητα γιατί εξίσου επικίνδυνα είναι με τα υπόλοιπα. Το βασικό μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από τι τροπολογίε μου είναι το εξή. Θα ήθελα να κατοχυρώσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση επιπρόσθετη σε σχέση με την διάθεση των αποβλήτων σε βαθύτερα γεωλογικά στρώματα. Δηλαδή μία ανακτήσιμα, ε, μία ανακτήσιμα γίνονται τα απόβλητα εφόσον ακολουθεί αυτή ακολουθηθεί αυτή η μέθοδος και θα ήθελα τα κράτη-μέλη να έχουν μια αναλλακτική μέθοδο. Όσα κράτη-μέλη το επιθυμούν ε, θα μπορούσαν να υποφεληθούν από την προϊούσα έρευνα και επίσης ε, τα θέματα ασφαλείας μην ξεχνάμε ότι ενδέχεται να περιπλεχθούν πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε φανταστεί στην αρχή. Οπότε θα ήθελα να προσθέσουμε ένα ορισμό σχετικά με την τελική αποθήκευση. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα είτε για τη διάθεση είτε για το final storage, την τελική αποθήκευση που θα ορίζεται ως η διάθεση των ενεργών αποβλήτων σε βάθος όπου δεν προβλέπεται ανάκτησή τους αλλά να είναι εφικτή ανάκτηση αν τεθεί ζήτημα ασφαλείας διότι προς το παρόν δεν είναι σαφέστατες οι σχετικές διατάξεις. Επίσης θέλουμε μία ρήτρα sunset ε, για το συγκεκριμένο νομοθέτημα, μία ρήτρα εκπνοής αν θέλετε, διότι μετά από δεκαετία καλούνται τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν ε, τα προγράμματά τους και κατόπιν θα γίνει και αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε αν πούμε ότι αυτό θα διαρκέσει μόνο 15 χρόνια, δίνεται έτσι η ευκαιρία να αναθεωρηθεί η πολιτική και να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη και οι έσκατες ε, τεχνολογικές εξελίξεις. σχετικά με την διάθεση των αποβλήτων σε βαθιά γεωλογικά στρώματα, πιστεύω ότι είναι ε, ε, πιο σόφρο να διατηρούμε την αλλακτική λύση της τελικής αποθήκευσης, ε, δηλαδή τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν να έχουν αυτή την επιπρόσθετη λύση της τελικής αποθήκευσης σε σχέση με την ε, διάθεσή τους ε, σε βαθιά γεωλογικά στρώματα. Ε, τα κράτη-μέλη τους έλους θα πρέπει να μας προτείνουν, να μας παρουσιάσουν την τελική τους λύση σε εισαγωγικά για την διάθεση των αποβλήτων στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος. Ο στόχος είναι να μην έχουμε τα απόβλητα μέσα στη φύση ΕΣΑΗ e και να μην έχει ληφθεί καμία απόφαση σε σχέση με την τύχη αυτών των αποβλήτων τέλος. Um, σχετικά με την εξαγωγή των αποβλήτων ναι, και τα ε, λοιπά επιμέρους στοιχεία, νομίζω ότι είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να καταλήξουν συμφωνία σχετικά με μια υποδομή διάθεσης, ε, ε, ένα κέντρο διάθεσης. ένα κοινό κέντρο διάθεσης, αλλά ε, δεν νομίζω ότι επαρκούν οι διατάξει που ισχύουν για να εξαγάγουμε τέτοια απόβλητα. Δεν είμαστε ουδόλω σε θέση να ελέγξουμε το ποιε ευεξεργασία την χάνουν τα απόβλητα με το που ε, βγουν από την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και αυτό όμω είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε να στέλνουμε τα απόβλητα σε χώρε, σε μέρη όπου δεν μπορούμε να ελέγξουμε την τελική του διάθεση. Σα ευχαριστούμε, κ. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Να πω επίσης πως η συζήτηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη, αλλά ευαισθητώση είναι απαραίτητη προκειμένου να καταλήξουν σε κάποιους κανόνες. Χαίρομαι που μπορέσαμε να βρούμε μια διατύπωση η οποία μας ε, προτείνει κάποιες ε, λύσεις στο ε, πρόβλημα, όπως αναφέρει και η συνάδελφος, συνεργασία σε επίπεδο κρατών μελών, κοινέ εγκαταστάσεις αποθήκευσης, κοινή χώρα αποθήκευσης ή και σε περιπτώσεις εξαγωγής των ραδιενεργών αποβλήτων ή του αναλωμένου υλικού, λιμενικού Χρειάζεται όμως ε, να, έχουν, να υπάρχουν πλήρη φάκελοι σχετικά με το περιεχόμενο των ε, αποστολών. Είμαι πεπισμένη και είμαι πεπισμένος μάλλον και ξέρω ότι η συγκεκριά του έλαβε υπόψη της ε, το θέμα αυτό ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να περιπλέξουμε έτσι περαιτέρω τα πράγματα και τις ε, ρυθμίσεις για να μην δημιουργήσουμε έναν πολύ άκαμπτο ε, μηχανισμό διοικητικό, διότι ένας ε, ιδιαίτερα περίπλοκος και άκαπτος διοικητικός μηχανισμός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα διαφάνειας και ενημέρωσης του κοινού. Αν λοιπόν η όλη διαδικασία είναι περίπλοκη, πολλές φορές αυτό αποβαίνει εις βάρος ε, της διαφάνειας για την διαχείριση αυτών των ραδιολογικών υποβλήτων και των αναλωμένων καυσίμων και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Θεωρώ ότι η συζήτηση επί της εκθέσεως ήταν ε, όντως δύσκολη αλλά βοήθησε αναφίβολα στο να βελτιωθεί περαιτέρω η έκθεση και εξ ονόματος ε, της πολιτικής μου ομάδας μπορώ να πω ότι ορισμένε πτυχέ επιλήθηκαν πολύ σωστά από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χέρτσοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήδη συζητήσαμε το θέμα και είδαμε πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο πλαίσιο των πολιτικών ομάδων χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι αυτές οι διστάμενες απόψεις υπάρχουν αλλά ταυτόχρονα υπάρχει συνένεση μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων πως ανεξάρτητα με τα όσα συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν ίσως ακριβώς και γι' αυτό το λόγο στη διαχείριση των ραδιοεργών αποβλήτων πρέπει να υπάρξει πρόοδος. Γι' αυτό λοιπόν δεχόμαστε την πρόοδο την οποία έχει επιτύχει και το Συμβούλιο σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε εξάλλου και το Συμβούλιο για τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια της ε, εκπόνησης της εκθέσεως, διότι σε ό,τι φορά την οδηγία αυτή, εμείς βασιζόμαστε στην εφαρμογή της συνθήκης της ε, Euratom και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά και πριν από την υποβολή των τροπολογιών, το Συμβούλιο έδειξε ότι ήταν διατεθειμένο να ακούσει την άποψη του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα τη συνεργασία. Υπάρχει και εδώ εκπρόσωπο τη Ουγγρική Προεδρία. Πρέπει λοιπόν να καταγράψουμε την πρόοδο που έχει ήδη Φυσικά αυτό δεν επαρκεί. Χρειάζεται παράλληλα να συμμορφωθούμε προ ε, τη νέα κατάσταση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη χρηματοδότηση. Απαιτείται να εξεύρουμε την λύση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η βιομηχανία και να υπάρχει ένας μακροχρόνιος προγραμματισμός. Ε, προς αυτή την κατεύθυνση κατεύθυνσαν αρκετές τροπολογίες και πιστεύω ότι θα καταληθούν κι άλλες. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση αναφορικά με τα εθνικά προγράμματα και τονίζω πως υπάρχει ήδη μια ικανοποιητική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Να πω κάτι πια πράγματα τα οποία ήδη έθιξαν οι προαλήσαντες συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά το safety case, κατά διάρκεια της κατάρτισης οδηγίας αναφορικά με την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, όλοι θεωρούσαν ότι η μεταφορά της οδηγίας για τα ραδιενεργά απόβλητα θα γινόταν δίχως ε, προσκόμματα, δίχως εμπλοκές ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θέσει σε αυτήν την οδηγία τα θέματα ασφαλείας. Εν τω μεταξύ υπήρξαν ε, σημαντικές αλλαγές διότι έγιναν κάποιες δοκιμές, κάποια stress test και προέκυψε ότι χρειαζόταν να τροποποιηθεί η οδηγία αναφορικά με την ε, διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων. Ως εκ τούτου οι παράγραφοι που αφορούσαν την πυρηνική ασφάλεια χρειάζεται να τροποποιηθούν Λοιπόν, παράλληλα με την τροποποίηση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια είναι εύλογο να ε, συμπεριληφθούν τροποποιημένες αυτές οι παράγραφοι αλλά αναφίβολα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και πολλέ τροπολογίε κατά την άποψή μου θα κατατεθούν περί αυτών των παραγράφων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό και βέβαια πω και εδώ θα κατατεθούν τροπολογίε. Και αναφέρομαι στο ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την διάθεση αυτών των αποβλήτων. Φυσικά δεν μπορεί να ε, έχει το μονοπόλιο, δεν μπορεί να περιοριστεί λοιπόν ο ανταγωνισμό σε αυτόν τον τομέα. Άρα χρειάζεται να επιβάλλουμε στους ε, φορείς ε, οι οποίοι χειρίζονται τα πυρηνικά απόβλητα το ότι οι ποσότητες χρειάζεται να ελαχιστοποιηθούν ε, ε, η ραδιενέργεια θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλή και οι επιχειρήσει που ασχολούνται με την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων φυσικά ενδιαφέρονται για ποσότητε ιδιαίτερα υψηλέ σύμφωνα με κάποια οικονομικά πρότυπα με τα οποία λειτουργούν. Αλλά η ραδιενέργεια θα πρέπει να είναι χαμηλότερη δυνατόν προκειμένου να εγγυηθούν με την καλύτερη δυνατή ασφάλεια. Και εδώ θα καταθέσουμε τροπολογίες. Η συγγήτρια έλαβε υπόψη τη ε, και μια άλλη πτυχή του προβλήματο, ε, δηλαδή στην ε, μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται οι νέοι οι νέες επιχειρήσεις ε, που εισέρχονται στην αγορά. οποιοςδήποτε λοιπόν, ε, οποιαδήποτε επιχείρηση που ασχολείται με την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτήν την δραστηριότητα και εδώ περνάω στο θέμα της εισαγωγής και εξαγωγής αποβλήτων πρόεδρος ε, Σασέτα έχει, συγγνώμη, ο επίτροπος ε, Σασέτα έχει μια συγκεκριμένη θέση πάνω στο σύστημα αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ε, προκαλέσουμε την δημιουργία μονοπωλίων στον τομέα αυτών. Θεωρούμε λοιπόν πως αν και στην φίλοι υπάρχουν λίγοι χώροι εναπόθεσης αυτών των αποβλήτων, εμείς δεν μπορούμε να περιορίσουμε τις Εξαγωγέ ε, διότι και τι εισαγωγέ. Είμαστε ιδιαίτερα ελαστικοί ε, σε αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν ε, αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Εξόμενος λοιπόν της πολιτικής μου ομάδας θέλω να πω ότι συμφωνούμε με την άποψη του Συμβουλίου και άρα με την άποψη της ε, Κομισιόν, με τις ε, σε σχέση με την αρχική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, χρειάζεται λοιπόν να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας έγκαιρα και θέλω να το τονίσω το έγκαιρα διότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό η έκθεση να εγκριθεί εγκαίρως πριν από την ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου. Εμεί ω ομάδα παρουσιάσουμε διατηρημένη το πράξη. Ευχαριστώ. Ε, προτείνω να χρησιμοποιήσουμε από εδώ και μπρο ένα όριο δύο λεπτών, αλλιώ δεν θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, ο κύριο Μπιουτικόφερ τώρα από του υπόλοιπου συναδέλφου. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν μου αρκούν δύο λεπτά. Και δεν ξέρω και αν είναι και σωστό αυτό. Μα κύριε Μπουτικόφερ για να το ξεκαθαρίσω. Άφησα να μιλήσουν λίγο περισσότερο οι προλαλήσαντες γιατί ήταν οι ισχυώδεις εισηγητές. Εντάξει, τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά παρακαλώ, εάν νομίζω ο καθένας περιοριστεί λίγο, θα τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσω, λέει ο κ. Σπιτικόφερ. Οπότε φεύγουν οι έπαινοι και θα πω, θα ασκήσω κυρίως ε, κριτική. Και φταίτε εσείς κύριε Πρόεδρε άρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο ορισμός των πυρηνικών αποβλήτων. Κατά την απόψή μας, ο ορισμός που προτείνεται εδώ πέρα είναι πολύ ήπιος. Ήτανε μεγάλη συζήτηση για το πόσο θα πρέπει να κάνουμε εικασίες για μελλοντικές ε, λύσεις, τεχνικές, ε, το εάν θα πούμε προβλέπετε ή κάποιο άλλο ρήμα ή envisaged. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι παραθυράκια, δηλαδή το τι φαντάζεται ο καθένας και εγώ αν έχω φαντασία μπορώ να φαντάζομαι ε, ότι θα γίνουν διάφορα πράγματα στο μέλλον και άρα α, ξεφεύγουμε από τον ορισμό των αποβλήτων. Δεν είναι έξυπνο αυτό. Επίσης δεν θεωρούμε πως το, η εξόριξη και τα απόβλητα της εξόριξης ουρανίου πρέπει να εξαιρεθούν. Υπάρχουν και πυρηνικά απόβλητα τα οποία προκύπτουν από την εξόριξη σπανίων γεών και άλλα πράγματα που δεν καλύπτονται από τους ορισμούς. Πρώτον αυτών. Είναι δηλαδή πολύ ήπιοι ορισμοί δεύτερον. Το παράθυρο που ανοίγει εδώ πέρα για εξαγωγές, το βρίσκω αυτό εντυπωσιακό. Δηλαδή λέτε πως εάν ε, βάλουμε περιορισμούς θα δημιουργήσουμε μονοπόλια. Εάν όμως οι περιορισμοί έχουν τόσες τρύπε ε, σε έχει αυτό εδώ πέρα, τότε δημιουργούμε ζώνες ε, ανασφάλειας. Δείτε μόνο τι έγινε στο Μαγιάκ στη Ρωσία για να διαπιστώσουμε ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με την εξαγωγή πυρηνικών αποβλήτων από την Ένωση. Συμφωνώ πλήρω με την κυρία Χολ. Πρέπει τουλάχιστον να φροντίσουμε τα απόβλητα που παράγουμε στην Ένωση να αποθηκεύονται στην Ένωση εάν όχι ε, στη χώρα που έχει την ευθύνη, γιατί τα έχει χρησιμοποιήσει κιόλα. Ο κύριος συνάδελφος λέει πως θέλει να εμποδίσει την εξαγωγή. Ο κύριος Επίτροπος και αυτό ήταν βασικό ε, σημείο της Κομισιόν. Γιατί ήταν έξυπνο αυτό και λυπούμε για το ότι προσπαθεί ε, να το ανατρέψει η Επιτροπή μας. Και τρίτον και τελευταίον κύριε Πρόεδρε, έχω κάποιες δυσκολίες με τον ορισμό αυτόν εδώ πέρα της αναστρεψιμότητας. Στη Γερμανία, στην περίπτωση του ΆΣΕ, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η αρχή της αναστρεψιμότητας. Αλλά εάν βλέπετε πόσο ο ορισμός επιτρέπει κάποια κράτη-μέλη να αφήνουν ανοιχτό τον αποθηκευτικό χώρο και αυτό είναι άρα εγγύηση αναστρεψιμότητας, ε, τότε είναι πάρα πολύ χαμηλό, χαμηλός ο πύχης, γιατί είναι ε, τεράστιο το κόστος μετά της ε, ανάκτησης και δεν είναι σωστό να έχουμε πάλι τόσο ήπιο ορισμό. Οπότε, αν και χαιρόμαστε για κάποια σημεία, όπως στην αρχή ο πληρώνει ή και τα στρατιωτικά απόβλητα, έχουμε κάποια σημεία στα οποία πιστεύουμε πως δεν ανταποκρινόμαστε ε, στις ανάγκες με τα κριτήρια αυτά που πρότεινε δηλαδή ο κύριος Σέτιγκερ δηλαδή η ε, καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και επιστήμη. Ευχαριστώ. Ενέν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο λεπτά. στις κοινότητες και στους δήμους των χωρών μας αποφασίσαμε σχετικά με την διάθεση των ε, οικιακών ε, αποβλήτων σε κοντινές ε, περιοχές, χώρους, κοντά στις χώρες του οποίου παράγονται. Και είναι και φυσιολογικό να μας ζητήσουν να αποφασίσουμε και για τα πυρηνικά απόβλητα, απόβλητα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή στο πιο κοντά στο χώρο παραγωγής τους. Και θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν σε αυτούς που παρήγαγαν τα απόβλητα να αναλάβουν τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Αυτό νομίζω είναι προφανές. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα ασχοληθούν. Να πάρουμε την περίπτωση της Γαλλίας, της χώρας μου. Παλιά είχαμε την παραγωγή της ενέργειας στο πλαίσιο μιας δημόσιας υπηρεσίας και όλες οι επιχειρήσεις ε, ε, επωφελήθηκαν από την παραγωγή αυτού του ηλεκτρικού ρεύματο κλπ. κλπ. Έτσι λοιπόν το, υπήρχαν λοιπόν ε, πολλά ε, θετικά αποτελέσματα και από την πυρηνική ενέργεια αλλά και πριν από λίγο καιρό μας είπαν ότι θα πρέπει να έχουμε δύο μόνο επιχειρήσεις ε, στον τομέα της ενέργειας και όχι παραπάνω. Μία έχουμε τη ΔΕΗ της Γαλλίας και την ΖΕΝΤΕΕΦ την οποία ανήκει σε ιδιωτικά κεφάλαια. Πώς θα πρέπει να κάνουμε τώρα για να υπάρχει η η κατανομή του κόστους ε, με τρόπο δίκαιο, διότι όλοι υποφελήθηκαν από την κατάσταση αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αφήσουμε ελεύθερη τα κράτη-μέλη που έλαβαν τέτοιου είδου αποφάσεις να διαχειριστούν με ευθύ τρόπο τόσο για σήμερα όσο και για το αύριο την ε, ανάγκη ε, ε αγγίησης απόλυτης ασφάλειας για τους πολίτες και αν είναι απαραίτητο να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις από χώρα σε χώρα Κάποιε οργανώσεις μάλλον ε, κοινέ, τότε θα πρέπει να ελέγχονται. Τώρα σε ό,τι φορά τα μονοπόλια να σα υπενθυμίσω πως ε, με το πρόσχημα τη απελευθέρωση φιλελευθερωποίηση κλπ. Ε, συχνά στην Αφρική βρίσκουμε πυρηνικά απόβλητα που έχουν ταφεί, βρίσκουμε καράβια τα οποία βυθίζονται στην θάλασσα απλά και μόνο επειδή απελευθερωποιήσαμε και επιτρέψαμε σε επιχειρηματίες ε, να κερδοσκοπήσουν εις βάρος της ασφαλείας μας. Ευχαριστώ, Βιδάλκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Τζόρνταν για την εξαίρετη εργασία της. Είναι γεγονός ότι υπό το φως των γεγονότων της Φουκουσίμα το σενάριο έχει αλλάξει άρδιν, αλλά η ανάγκη για αυτήν την οδηγία είναι πράγματι επιτακτική. Έχουμε διαφορετικές θέσεις, διστάμενες απόψεις στην, στο κοινοβούλιο μας αναφορικά με το ενεργειακό μείγμα και ήταν δύσκολο λοιπόν να υιοθετήσουμε κάποιο ψήφισμα για το θέμα της Φουκουσίμα στην τελευταία σύνοδο αλλά τα πυρνικά απόβλητα βρίσκονται εδώ και υπάρχει ευθύνη την οποία πρέπει να φέρουμε και ευθύνε που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υποστηρίζω τι τροπολογίε τη κυρία Τζόρνταν, την προσπάθειά τη για μεγαλύτερη διαφάνεια, την πρότασή τη ε, για την, ε, την υποχρέωση των ε, εξοδοτημένων αρχών να αναφέρουν στις ε, ρυθμιστικές αρχές ε, το ζήτημα της ασφάλειας, ε, το θέμα της αναγνώρισης της σημασίας της έρευνας στον τομέα της ελληνικής ενέργειας αλλά και το ζήτημα της αρχής της ρευσιμότητας και τονίζει επίσης τον ρόλο της των εθνικών, των ρυθμιστικών, εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Υπάρχει ένα σημείο Συμφωνώ για το ζήτημα των χώρων ε, αποθήκευσης. Ε, αυτά μπορούσαμε να συζητήσουμε όμως κυρία Τζόρνταν το, κάποιο, επίπεδο των λεπτομεριών ε, που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κανονισμό. Αλλά συμφωνώ ότι διασφαλίζοντας ε, τις βασικές αρχές ε, είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Και υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο θα διαφοροποιηθώ με την άδειά σας ε, κυρία Τζόρνταν. Έχω διαφορετική άποψη από εσά. Μιλάμε για το άρθρο σχετικό με την χρηματοδότηση το σημαντικό, κυρία Τζόρταν, είναι τα χρήματα να υπάρχουν και να είναι διαθέσιμα όταν και εφόσον χρειαστούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ενθυμίστε πως ε, η προσπάθεια που κάναμε το 2004 απέτυχε ακριβώς λόγω του ότι ζητήσαμε πάρα πολλά από το Συμβούλιο και το πράγμα δεν προχώρησε. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν είναι πιο προσεκτική, αλλά όχι λιγότερο αποτελεσματική. Συμφωνώ λοιπόν με το να στηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν και όχι την δική σας στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ όμως για την εξαιρετική σας εργασία και προσβλέπω στην επικείμενη συζήτηση. Ευχαριστώ. Yes, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τη Ρωμάνα για τη δουλειά της. Και θα επικεντρωθώ σε ένα ζήτημα. Θα ήθελα να εκφράσω τις ανησυχίες μου για τις ε, πιθανές δυσκολίες για την εφαρμογή του άρθρου 4.3 απέτηση διάθεσης ε, όλων των αποβλήτων στην επικράτεια της Ένωσης. Η αναζήτηση λύσεων εντός της Ένωσης μόνο είναι πολύ περιοριστική και μπορεί να, δώσει, να προκαλέσει και νομικά και κοινωνικό οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι σαφές πώς ε, ωφελείται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αυστηρή απαγόρευση διάθεσης σε τρίτες χώρες. Πρώτα απ' όλα, το άρθρο αυτό θα μπορούσε να θέσει την εφαρμογή μακροχρόνιων συμβολέων που έχουν κλείσει κάποια κράτη-μέλη με τρίτες χώρες. Συμβάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρατόμ και την υπηρεσία προμήθειας καυσίμων. Δεύτερον, το άρθρο αυτό στην πράξη καθιστά δυνατές ε, τις περιφερειακές και παγκόσμιες λύσεις και αμφισβητεί τις εφαρμογές ε, υφιστάμενων πρωτοβουλειών π.χ. την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Μείωση των Απειλών, όπου, χώρες, όπου συμμετέχουν χώρες ε, εκτός Ένωσης με την απαγόρευση αυτή. Προσπαθούμε επίσης να απομονώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις γειτονικέ χώρες, από παγκόσμιες και περιφερειακές λύσεις, ενώ πρέπει να συμβεί ακριβώ το αντίθετο. Να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία για να επιτύχουμε καλύτερη παγκόσμια ασφάλεια. Όλοι γνωρίζουμε πως η πυρηνική ασφάλεια και η ραδιολογική ασφάλεια δεν έχει σύνορα. Το άρθρο αυτό επίσης δεν ε, στέκει και οικονομικά. Γεγονός είναι πως σε μικρές χώρες με πυρηνικά προγράμματα το οικονομικό βάρος ε, από την κατασκευή ε, εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων μπορεί να καταστήσει οικονομικά σύμφωνα την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού εργοστασίου. Γι' αυτό οι απαιτήσει αυτού του άρθρου εμποδίζουν την ε, ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό θέλουμε με αυτή την οδηγία. Είναι προφανές πως το σκεπτικό που υποκρύβεται εδώ πέρα και αφορά την απαγόρευση ουσιαστικά πρέπει να επανεξεταστεί. Κύριος Μπέλετς. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ, σβήστε. Thanks, uh, Chairman. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά όπως είπατε θα περιοριστώ σε δύο άρθρα, το 3 και το 10. Πρώτα απ' όλα το άρθρο 3 που αφορά τους ορισμούς, γιατί εκεί πέρα λέτε πως η ταφή είναι αποθήκευση πιθανώς οριστική. Αυτό θα οδηγήσει σε κάποια σύγχυση, γιατί το πιθανώς οριστική μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση πως ε, κάθε εγκατάσταση ταφής ε, θα πρέπει να είναι μια υπόγεια αποθήκευση που μπορεί να γίνει οριστική ε, αποθήκευση. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Αν υπάρχει μια τέτοια υποχρέωση ε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύσεις που θα είναι λιγότερο ασφαλείς από αυτές που έχουμε σήμερα. Ε, αυτό λοιπόν όσον αφορά τους ορισμούς. Δεύτερη παρατήρηση για το άρθρο 10 και τις σχετικές τροπολογίες της εισηγήτριας αφορά εδώ πέρα το θέμα το κόστος και τα μέσα που πρέπει να προβλέψουν τα κράτη-μέλη για να καλύψουν το κόστος. Και θα ήθελα να αναφερθώ εδώ πέρα στο κόστος που συνδέεται με την συντήρηση. Πράγματι μπορεί να έχει νόημα αυτό εδώ πέρα για μία εγκατάσταση διάθεσης που αποθηκεύει στην επιφάνεια αλλά όταν μιλάμε για ταφή σε βάθος μεγάλο, γεωλογικό, δεν ε, είναι τόσο προφανές. Ε, κάτι τέτοιο λένε οι ειδικοί, γιατί η ασφάλεια μιας υπόγειας αποθήκευσης ε, δεν σχετίζεται με τη συντήρηση. Ίσως συντήρηση λέμε πως θα πρέπει να υπάρχει κάποια επιτήρηση ίσως θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε εδώ πέρα. Και, εάν μου επιτρέπετε, μία τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, για την χρηματοδότηση και το κόστος. Οικονομικά μέσα σημαίνει πως ε, θα πρέπει να καλύπτεται η πτυχή της ε, πυρηνικής ασφάλειας. Ε, Εσύ το συμπεριλαμβάνετε αυτό ή, ή, ή όχι. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Äh, Έχουμε λοιπόν ε, γύρω στα 15 λεπτά γιατί μετά θα έρθει η κυρία Επίτροπος και θα ήθελα να ακούσω βεβαίως και τους εκπροσώπους ε, Κομισιόν και Συμβουλίου και την εισηγήτρια ξανά. Οπότε ε, να παρακαλέσω να το θυμάστε. Πρώτα απ' όλα να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν. Κύριος Φάρος, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψατε μου παρά την ε, πίεση του χρόνου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή έκθεση που υπέβαλε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία έτσι κάπως συνοπτικά. Το πρώτο η αναστρεψιμότητα. Δεν την αποκλείσαμε στην πρότασή μας την ε, αναστρεψιμότητα, την έχουμε ρητός αφήσει ανοιχτή, αλλά δεν ορίζουμε πως ε, θα πρέπει να είναι δυνατή υπό συγκεκριμένα κριτήρια. Θεωρούμε πως κάθε κράτος μέλος το οποίο θέλει να κάνει εγκατάσταση τελικής αποθήκευσης θα έχει τους δικούς του κανόνες αναστρεψιμότητας οι οποίοι διαφέρουν αυτή τη στιγμή. Οπότε, επαναλαμβάνω, δεν το αποκλείουμε, επαφίεται στα κράτη-μέλη να το ορίσουν. Οικονομικά μέσα. Ο κύριος Βιδάλ Κουάντρας στην παρέμβασή του κατέστησε σαφές ποιες ευαισθησίες κρύβονται πίσω από αυτό τον όρο. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διασφαλιστεί πως όταν θα χρειάζονται θα είναι διαθέσιμα τα μέσα για την κατασκευή ενός χώρου τελικής αποδίκευσης. Το... να πάμε τώρα ακόμη παραπέρα, το κάναμε αυτό σε μια σύσταση του 2006 και βλέπουμε πως εφαρμόζεται αυτή η σύσταση σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως το Κοινοβούλιο μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα και να θέσει περαιτέρω διατάξει στην ισχύ, μέσω της παρεμβασή μου θα ήθελα να τονίσω πως σημαντικό είναι να υπάρχουν τα λεφτά. Όχι να εφευρεθεί η διαδικασία πως θα είναι διαθέσιμα τα λεφτά. Και ένα πολιτικό θέμα μετά, απαγόρευση εξαγωγής για πυρηνικά απόβλητα. Κοιτάξτε, για να είμαστε σαφείς, πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα η διάκριση μεταξύ πυρηνικών αποβλήτων και άλλων ουσιών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Και ο κύριος Επίτροπος νομίζω σε πάρα πολλά σημεία επανέλαβε πως μόνο τότε υπάρχει εγγύηση ασφάλειας όταν μπορεί κανείς να επηρεάσει την ασφάλεια των αποθηκευτικών χώρων. Και αυτό γίνεται, είπε, όταν αυτοί οι χώροι είναι εντός της κοινότητας. Οπότε το συμπέρασμα το οποίο προέκυψε είναι πως επί της αρχής θα πρέπει να παραμένουν εντός κοινότητας τα απόβλητα για να μπορούμε να τα εξετάσουμε. Και το έχει πει Πολάκης. Ξέρω πως υπάρχει μια σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο, ξέρω πως θα υπάρξει μια συμβιβαστική πρόταση, αλλά θα την δούμε όταν προκύψει. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λέμε ως αρχή είναι πως εάν θέλουμε σίγουρη τελική αποθήκευση θα πρέπει να μπορούμε να την αποθηκεύσουμε γιατί σε κάποια τρίτα κράτη-μέλη δεν έχουμε καμία επιρροή ως κοινότητα. Μετά. Για τα υπόλοιπα σημεία βεβαίως θα δούμε τις εθνικές εκθέσεις. Βεβαίως η μελέτη ασφαλείας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής για να ε, δοθούν άδειες. Σε ένα σημείο υπάρχει μια παρεξήγηση και αυτό αφορά τον ορισμό του τελικού αποθηκευτικού χώρου. Αυτό το οποίο λέμε final storage, οι ειδικοί το θεωρούν αντίφαση. Disposal που λέμε στα αγγλικά, διάθεση, ε, ούτως ή άλλως υποκρύπτει την έννοια τελική. Όταν μιλάμε για αποθήκευση, μιλάμε για χρονικούς ορίζοντες που είναι στην καλύτερη περίπτωση 30 έτη και όταν μιλάμε για αποθήκευση μιλάμε για ενδιάμεση αποθήκευση. Μία, παρ... Ε, μία παράκληση θα είχα εδώ όσον αφορά το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την ενδιάμεση αποθήκευση βλέπουμε ήδη και αντλούμε διδάγματα από τη Φουκουσίμα. Ενδιάμεση αποθήκευση δεν είναι σίγουρη και διαρκής λύση. Ενδιάμεση αποθήκευση σημαίνει αποθήκευση χωρίς περιορισμό. Και χωρίς περιέκτη και ε, επειδή ε, ο χρόνος πιέζει όπως είπατε κύριε Πρόεδρε θα περιοριστώ σε αυτά και ε, δεν θα μπω σε άλλα σημεία. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις σας να δώσω στον ε, πρόσωπο του Συμβουλίου, τον κύριο Λάσλο Κομπλιγκέρ, τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρίε και κύριοι. Χαίρομαι που παρευρίσκομαι σήμερα στην συνεδρίασή σας και ευχαριστώ την Ρωμάνα Γιόρνταν Σίζα για τις ε, παρατηρήσεις της ε, και πράγματι μας έδωσε ε, πολύ έγκαιρα τα έγγραφα. Ήταν μια εμπειρία πολύ υποδομητική. Χαίρομαι που στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου μπορέσαμε να εργαστούμε παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την περασμένη Παρασκευή εξετάσαμε την τελευταία εκδοχή του κειμένου και σε αυτήν περιλαμβάνεται η αρχή της, της Επίση Επίσης υπάρχει μια σημαντική πτυχή της έρευνας και της ε, ανάπτυξης. Ε, λοιπόν, τα δύο όργανα λειτουργήσαν θα έλεγα με τρόπο παράλληλο. Θα ήθελα να ασχοληθώ τώρα με το θέμα των εισαγωγών-εξαγωγών. Ευθύ εξ αρχή η Ουγγρική Προεδρία τόνισε την σημασία των εγκαταστάσεων διάθεσης των ραδιοενεργών αποβλήτων και ελπίζω να μπορέσει να μπορεί να φέρουμε σε αίσιο πέρας και αυτή την οδηγία. Ε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να εκπονήσουμε ένα έγγραφο αποδεκτό από όλα τα κράτη-μέλη. Προ το παρόν ε, δουλεύουμε πάνω στι συμβαστικέ προτάσει που έχουν κατατεθεί σε όλη φορά τον περιορισμό τη απαγόρευση εξαγωγών. Δηλαδή, ε, από συγκεκριμένε προποθέσει θα μπορούμε να επιτρέπουμε τι εξαγωγέ αυτέ. Χρειάζεται λοιπόν να ξεβρεθούν κάποιε συμβαστικέ λύσει. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα επί δύο ακόμα ζητημάτων. Πολλοί βουλευτέ αναφέρθηκαν στην ε, φυσική καταστροφή στην Ιαπωνία που ακολούθησε, που ακολούθησε μετά η πυρηνική καταστροφή, η καταστροφή μάλλον του πυρηνικού εργοστασίου. Και θα ήθελα εδώ να κάνω μια παραμπομπή. Η οδηγία που αναφέρεται σε θέματα ε, ε, διάθεσης των αδιανογών απολύτων θα πρέπει να προωθείται στο μόνο δυνατόν. Οι λοιπόν στην Ιαπωνία επιτάχυναν τις ε, διαδικασίες. Ε, και μια τελευταία παρατήρηση το 2009 ε, εγκρίναμε την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια. Στην περίπτωση αυτή επρόκειτο για μια οδηγία πλαίσιο και υπήρχε η δυνατότητα για τις εθνικές αρχές να υιοθετήσουν άλλες ρυθμίσεις με πολύ πιο συγκεκριμένα επίπεδα Τώρα έχουμε φτάσει σε 200 επίπεδα αναφοράς, τα οποία έχουν ε, όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα και στην διάθεση των ραδιοενεργών αποβλήτων ε, χρειάζεται το συντομότερο δυνατόν να ε, αυτή η οδηγία προκειμένου να ε, πετύχουμε ένα σύστημα αναφοράς που θα ισχύσει όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ και θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Γιώργαν Σίσελ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ του συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Συμβούλιο για τα σχόλιά του. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες τις παρατηρήσεις και διαβλέπω περιθώρια συμβασμών, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία επί των οποίων υπάρχουν πιο σαφείς διαφωνίες, αλλά βέβαια θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε να εξεύρω μια κοινή θέση. Υπόθηκε ότι χρειάζεται να ε, χτενίσουμε κάπως ε, τις, ε, τους ορισμούς ναι, αναφίβολα θα λάβω υπόψη μου όλες τις παρατηρήσεις ε, που ζητούν ε, την ύπαρξη ενός υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας και μια αποτελεσματικότερη λειτουργία της ε, αγοράς. Δέχομαι επίσης και τις θέσεις που εκφράστηκαν αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται να εξεύρει λύσεις ε, οι οποίε ε, θα είναι λογικές αλλά και αποδεκτές προκειμένου να ληφθούμε σοβαρά υπόψη. Ε, Μπελέν ε, μου έκανε δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα της συντήρησης φυσικά όλες οι εγκαταστάσεις στις οποίες αφορά η οδηγία δεν ε, πρόκειται να γεμίσουν με απόβλητα και να ε, κλείσουν, θα λειτουργήσουν για ε, αρκετά χρόνια. Γι' αυτό έχω συμπεριλάβει και το κόστος συντήρησης. Επίσης υπάρχει ανάγκη ελέγχου και εποπτείας τώρα τα οικονομικά μέσα τα οποία απαιτείται να υπάρχουν ε, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ατυχήματος, ε, σοβαρού ατυχήματος. Κατά την άποψή μου αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της οδηγίας ε, αναφορικά με την πυρηνική ασφάλεια. Τώρα, σε ό,τι φορά την χρηματοδότηση, <coughs> γνωρίζω πως ε, υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίες ε, που πάνε πολύ πιο μακριά από τις προτάσεις Κομισιών και γνωρίζω ότι υπάρχει κίνδυνος το Συμβούλιο να μην δεχθεί αυτό το κείμενο, το κείμενο τροπολογιών ότι συνέβη το 2001-2003 όταν η οδηγία απορρίφθηκε αφού είχα συμπεριληφθεί κάποιες προϋποθέσεις χρηματοδότησης ιδιαίτερα αυστηρές ε, και απαιτητικέ ε, Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Συμφωνώ ότι χρειάζεται να πετύχουμε χρηματοδοτικούς πόρους ε, ικανοποιητικούς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους φόβους του πληθυσμού και των πολιτών μας. Εμείς τόσο πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια κοινή θέση όταν θα εξετάσουμε την τροπολογία για τη χρηματοδότηση. Τώρα, αναφορικά με τις ε, εξαγωγές, ακούστηκαν ε, ποικίλα σχόλια. Είμαι διατεθειμένη να συζητήσουμε για ε, την εξέβρεση μιας κοινή θέσης, μιας συνεντικής άποψης. Δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί. Το γνωρίζω από την σλοβενική εμπειρία. Έχουμε ένα πυρηνικό εργοστάσιο σε συνειδιοκτησία με τους Κροάτες γείτονες και η Κροατία χρειάζεται να ε, συμμετάσχει κατά το ίμιση στην διαχείριση των αποβλήτων. Μέσω τόσο καταλήγω ε, ευχαριστώντα ε, όλους του συναδέλφους, όπως επίσης την Κομισιόν και το Συμβούλιο και ελπίζω ότι θα κατορθώσουμε να ξέρουμε μια κοινή θέση. Ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Να υπενθυμίσω πως η προθεσμία άλλαξε και είναι 12 Απριλίου 12 η ώρα για τις τροπολογίες. Αυτό δεν σχετίζεται με εμά, αλλά με τους μεταφραστές που χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Οπότε έρχεται πιο νωρίς η προθεσμία. Μετά στις 5 Μαΐου θα ξανασυζητήσουμε το θέμα και 26 Μαΐου πιθανότατα θα λάβει απόφαση η Επιτροπή μας. Ολομέλεια δεύτερη του Ιουνίου για την οριστική απόφαση. Αυτά για αυτό το θέμα και άρα τελειώσαμε και σχεδόν ε, ακριβώς την ώρα μας περνάμε στο σημείο 4 αλλά δεν έχει έρθει κυρία Επίτροπος. Εμείς τα καταφέραμε αλλά μου λέει η γραμματεία ότι είναι θέμα δευτερολέπτων. Δεν έχει νόημα τώρα να περάσουμε σε άλλο θέμα τη ημερησίας διάταξη, Κάνουμε μια μικρή διακοπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω. Καλωσορίζω και την κυρία Νέλη Κρούς, αντιπρόεδρο της Επιτροπής και θα ήθελα να ακούσετε την κυρία Επίτροπο. Σας καλωσορίζω λοιπόν και σας δίνω αμέσως τον λόγο για να κάνετε μια εισαγωγή και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μέχρι τις 5 η ώρα. Λοιπόν, κυρία Κρούς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω βεβαίως επίγνωση του ότι είναι τιμή για μένα να παρευρίσκομαι στη σημερινή σας συνεδρίαση γιατί θα τροφοδοτήσετε το στοχασμό μου και το προβληματισμό μου για το μέλλον. What is at stake. Ταυτόχρονα θα δούμε ποια είναι τα διακυβεύματα, τι έχουμε ήδη πετύχει, τι σχεδιάζουμε για το μέλλον. Λογικό είναι λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να έχουμε και τη συμβολή του Κοινοβουλίου για το επόμενο τμήμα του ταξιδιού, ας το χαρακτηρίσω έτσι. Έχουμε ένα διαρκή διάλογο, είμαστε όλοι ανοιχτοί στο διάλογο και Ειδικότερα θα έλεγα ότι μετά την ευρεία διαβούλευση που έγινε στην αρχή της ε, θητείας ε, περάσαμε σε συγκεκριμένες δράσεις το Σεπτέμβριο, δηλαδή εγκρίθηκε το επωνομαζόμενο ευρυζωνικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενέχει το πρώτο πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος RSPP και την ε, σύσταση για την πρόσβαση νέας γενιάς, NGA. Παρακολουθώ ε, από κοντά τις τόσο σημαντικές εργασίες της Επιτροπής σας ε, και δεν το λέω για να σας ε, κολακεύσω αλλά η έκθεση της Επιτροπής σας κυρία Τζαβέλα σχετικά με την ευρυζωνική επικοινωνία έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι πολύ λογική αυτή η πρόταση του Κοινοβουλίου και ευθυγραμμίζεται με όλα τα υπόλοιπα που διαμείβονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας, τις προσπάθειες που κάνουμε, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο. Σχετικά με το πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι χρειάζεται μια αποτελεσματική χρήση του φάσματος. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο ούτω ώστε να είναι διαφοροποιημένη και ποικίλη χρήση του φάσματος, ενώ ταυτόχρονα θα βρούμε μια λύση για τον αυξανόμενο όγκο το... της ασύρματης κυκλοφορίας δεδομένων. Πολλά διακυβεύονται, υπάρχουν πολλές προσδοκίες. Κάθε τρεις μήνες παίρνουμε νέα στοιχεία, κάνουμε νέες προβλέψεις. Ε, οι εξελίξεις είναι εντυπωσιακέ. Ε, ε, Όλοι μαζί, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρούμε εφαρμόσιμες συμβαστικές λύσεις επί της ουσίας και αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί εύκολα. Ε, δεν μας περιμένει ο χρόνος, ε, ο, σημειώνονται ραγδαίες εξελίξεις στον κόσμο και κανείς δεν θα περιμένει την Ευρώπη και θέλω να το τονίσω αυτό. Αύριο η Επιτροπή θα ψηφίσει και αυτό είναι ένα σημαντικότατο βήμα στην διαδικασία και ειλικρινά ελπίζω ε, στη συνεργασία με το Συμβούλιο τελικά να εγκριθεί η πράξη στη δεύτερη ανάγνωση. Το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται προφανώς ε, την σημασία του ραδιοφάσματος για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές ε, και για την ε, πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα όλες τις προκλήσεις αλλά κυρίως να είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο για την κυβερνό ασφάλεια τώρα Έχουν σημειωθεί πολλές ε, κυβερνοεπιθέσεις ε, κατά ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αυτό καταδεικνύει την ανάγκη που υπάρχει να συσταθεί μια ομάδα άμεσης ε, δράσης για την κυβερνοασφάλεια και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Μάρο Σεύκοβιτς, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και την υποφαινομένη, συμφωνήσαμε ε, από την 1η Ιουνίου να αρχίσει να λειτουργεί μια ομάδα προδιαμόρφωσης ε, ΣΕΡΤ, αυτή η ομάδα μια ομαδα σε σερτ αυτη δράσης ε, για τους υπολογιστές, και θα μπει σε πλήρως λειτουργική φάση το 2012. Δεν χρειάζεται να μακρηγορώ για να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα τρία θεσμικά ε, όργανα και συνεργασία για να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα από το 2012. Το Κοινοβούλιο προσφέρει επιρογνώμονες ε, για να συνδράμει στην όλη προσπάθεια. Επίσης, χρειάζεται να εργαστούμε περαιτέρω για το, την αρχή ΕΝΙΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων ε, και Πλήρων πληροφόριων ε, χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί εγκρίθηκε η πρόταση για παράταση της τωρινής θητείας ε, ως έχει για άλλους 18 μήνες ε, και είμαι ε, αισιόδοξη σε σχέση με την έγκριση της πρότασης από το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να περατωθεί η νομοθετική διαδικασία για την έγκριση της νομοθετικής πράξης για το ΕΝΙΣΑ το ταχύτερο δυνατόν. Πάντως είμαι αισιόδοξη και θεωρώ ότι ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε την πρώτη ανάγνωση της πράξης το Νοέμβριο. Ε, τώρα, για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία. Ε, στη, 31η Μαρτίου εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην Ουγγαρία αυτή τη βδομάδα θα έχουμε μια διπουργική διάσκεψη για το θέμα αυτό που με ιδιαίτερη βαρύτητα και για τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια δεδομένα δεν χρειάζεται να σε εξηγήσω τη σημασία ε, που έχει η κυβερνοασφάλεια στην παγκόσμια σκηνή. Πλέον ε, δεν είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Επίσης ε, συμμετέχουμε σε εργασίες, ομάδας εργασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙΠΑ για την κυβερνοασφάλεια και το κυβερνοέγκλημα που συγκροτήθηκε μετά τη Σύνοδο της Λισαμονός το 2010 και θα συνεχίσει να εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε το διαδίκτυο και την σταθερότητά του στο επερχόμενο IGF Forum, δηλαδή Forum για τη διαχείριση του ίντερνετ στο Ναϊρόμπι, όπου θα συμμετάσχει το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, το, ο στόχο μα, ο απότερο στόχο μα είναι όλοι να συμμετάσχουν, τα κράτη-μέλη, ο ιδιωτικό τομέα, η κοινωνία των πολιτών και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έχοντα μια αυξημένη εμπιστοσύνη, σχέση εμπιστοσύνη ανάμεσα στου χρήστες και στους πολιτέ ε, στο διαδίκτυο. Αυτό είναι απαραίτητο για, για να είναι πιο αποτελεσματικέ οι ε, επιγραμμικέ ε, συνδιαλλαγέ. Αυτό φυσικά δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, Εργάζομαι σε στενή συνεργασία με την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ σχετικά με την ανθεώρηση για την προστασία των δεδομένων και επίσης επεξεργάζομαι την απόφαση σχετικά με την ε, οδηγία για τα, την, τα απόρριτα στοιχεία στο διαδίκτυο που θα αρχίσει να ισχύει το Μάιο. Τώρα, τι ποια εργαλεία αυτορύθμισης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη σύμφωνη γνώμη και των ε, λεγόμενων cookies. Έχουμε κάνει δύο στρογγυλές τράπεζες και τώρα επιοτιμούμε τι προτάσεις του για να δούμε αν είναι επαρκή ή αν χρειάζεται κάποια επιπρόσθετη δράση. Ε, μπορεί να χρειάζεται ισχυρότερη δράση. Το 2010 επίσης προώθησε ένα στενό διάλογο ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ε, και να διαβουλεύσει για τις καθολικές υπηρεσίες, την ε, επιγραμμική ουδετερότητα και την ε, περιαγωγή σας ε, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στην Επιτροπή Ήτρε για την σημαντική συμβολή της ε, στην ε, κοινή σύνοδο Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιγραμμική ουδετερότητα. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τις αρχές του ανοιχτού ίντερνετ, του ανοιχτού διαδικτύου, της καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπουμε την αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών για την περιαγωγή. Μέχρι την 30 Ιουνίου θα καταθέσουμε νέες προτάσεις ε, και Σχετικά με το γραφείο, την ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Τηλεπικοινωνίες, ε, γνωστή με το ακρονίμιο BEREC, ε, θα προωθήσουμε διαφανέστερες νομοθετικές πράξεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, σχετικά με την μεταφορά ε, των ευρωπαϊκών νομικών πράξεων στα κράτη-μέλη, για το πακέτο το τηλεπικοινωνιακό να ξέρετε ότι είμαστε, σοβαρολογούμε μάλλον για την 26η Μαΐου και δεν θα διστάσουμε να εκκινήσουμε διαδικασία διαδικασίε αν χρειαστεί, αν δεν γίνει σωστά η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Για την ε, διάσκεψη ICT 2010 που έλαβε χώρα στι ε, Βρυξέλλες τον περασμένο Σεπτέμβριο, μην ξεχνάτε ότι μας περιμένει μια ακόμη σημαντικότερη χρονιά, διότι εξήγηλα ήδη ένα πακέτο πρόταση υποβολής προσφορών ε, της τάξης των 780 εκατομμυρίων ευρώ, που ανήκει στο ευρύτερο πρόγραμμα εργασίας, ε, δηλαδή έχουν ε, προβλεφθεί στο διαγωνισμό 1,2 δις και νομίζω ότι αυτό θα μας ε, βοηθήσει ώστε να προωθήσουμε τις ε, ε, πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό και να διευρύνουμε τα ωφέλη των νέων τεχνολογιών για ολόκληρη την κοινωνία. για να υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή όλων στην κοινωνία, αυξάνοντας ε, την προσβασιμότητα στο δίκτυο και προωθώντας την ενεργό και υγιή ε, γύρανση. Ε, τον περασμένο Νοέμβριο έγινε μία παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της προσβάσιμης ψηφιακής τηλεόρασης ADT για άτομα με περιορισμένες ανάγκες ή με αναπηρίες, χάρη στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σε πληροφορίε και να χρησιμοποιούν πλήρως την ψηφιακή τηλεόραση και με τον συνάδελφο Τζον Ντέλ τον Νοέμβριο δρομολογήσαμε το πρώτο, ε, την πρώτη πιλωτική εταιρική σχέση για την καινοτομία σχετικά με την ε, υγιή και ενεργό γύρανση Και με τις κοινέ μας προσπάθειες σύντομα ελπίζουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Επίσης ε, θέλουμε οι οικιακές υπηρεσίες ε, να παραμένουν σε χαμηλή τιμή και να είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, επίσης, στις 15 Δεκεμβρίου 2010 εγκρίναμε το σχέδιο δράσης ηλεκτρονικής κυβέρνησης, ούτως ώστε οι πολίτες και οι εταιρείες να χρησιμοποιούν πραγματικά την ενιαία αγορά και οι δημόσιες υπηρεσίες επίσης να είναι στα ακροδά δάκτυλα αν θέλετε, των πολιτών και των ε, επιχειρήσεων. Ε, η δέσμευση που έχουμε αναλάβει μέσα από πιλωτικά προγράμματα όπως ε, ηλεκτρονικές και κρατικές προμήθειες, ηλεκτρονική αναγνώριση και πλαίσιο διαλειτουργικότητας ε, αποσκοπούν στο να είναι πιο ευέλικτος ευρωπαϊκός δημόσιος τομέας. Αρχίζουμε να προετοιμάζουμε το διάδοχο του προγράμματος πλαισίου 7, δεν έχουμε φτάσει ακόμη και ο νέος όρος είναι κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Θα διαρευνήσουμε πολλές εναλλακτικέ λύσεις στην συνέλευση για την ψηφιακή ατζέντα που θα λάβει η χώρα εδώ στις Βρυξέλλες 16 και 17 Ιουνίου. Ευελπιστώ ότι θα είναι αθρώα η προσέλευσή σας γιατί είναι ε, το πρώτο μείζον γεγονός αν θέλετε στην ε, υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντα, του ψηφιακού θεματολογίου. Σας διαβεβαιώ ότι θα είναι συγκλονιστικά ενδιαφέρουσα η διάσκεψη αυτή. Ε, αν θέλετε μπορείτε να, ήδη να δηλώσετε υποψηφιότητα και θα δούμε, θα, είμαι σίγουρη ότι θα προκύψει ένας μακρύς κατάλογος αποδράσεις ε, για το μέλλον. Τώρα, τον Ιούνιο του 2010 πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιγράψει διάφορες διαστάσεις του διαδικτύου των πραγμάτων, όπως ε, ονομάζεται. Ε, δηλαδή, έχει δώσει το στίγμα του το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να αρχίσει μια πραγματική μελέτη για τη χρήση του διαδικτύου σε τομείς όπως προσωπικά δεδομένα, υγεία και είδαμε την περασμένη εβδομάδα ότι συμπεγράφει μια παγκόσμια ε, ε, σημασία συμφωνία για τις ε, ετικέτες ραδιοσυγνικής αναγνώρισης και Χαίρομαι πάρα πολύ διότι όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία έχουν αναδειχθεί πλέον σε προτεραιότητα και έτσι ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι αυτή, αυτό το ψηφιακό θεματολόγιο έχει κάποιο νόημα για τον ίδιο και για τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι το ότι συνιστά προτεραιότητα αυτό στην πράξη για την ενιαία αγορά δεν επαρκεί και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μπαρνιέ, θα πάρει τη σκητάλη και θα προωθήσει το θέμα. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων ε, και όχι μόνο. Και το βασικότερο είναι η εμπιστοσύνη που νιώθουν και οι πολίτες και ο υπόλοιπος κόσμος ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κατόπιν ε, ε, επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Τρει είναι οι στόχοι μα. Πρώτον, αναθεώρηση της οδηγία 2003 το 2012, δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους τους δημόσιους φορείς και νέες εφαρμογές για χρήση των δεδομένων του δημοσίου τομέα, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι κωδικοποίηση εκδηλώσεων που έγιναν σε πέντε διαφορετικές πόλεις, ούτως ώστε να εκμεταλλευόμαστε τα δεδομένα Eurostat ε, και όπως προβλέπεται στην ε, ψηφιακή ατζέντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διευρύνει τα ωφέλη της διαλειτουργικότητας, ε, την θέσπιση μιας κοινών προτύπων και το 2012 θα εξετάσουμε την πιθανότητα ανάληψης μέτρων, τόσο ώστε να έχουμε κοινά δεδομένα ασθενών και διαλειτουργικότητα των μητρών, στα οποία θα έχουμε ηλεκτρονικά πρόσβαση από όλα τα κράτη-μέλη. Ένα τελευταίο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος, ε, το cloud computing για το 2012. Το σημαντικό είναι να επικρατεί η διαφάνεια και η διαβούλευση θα αρχίσει σε λίγες εβδομάδες. Ε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σχετικά με αυτό το ζήτημα και ελπίζω να τροφοδοτήσετε και εσείς τις εργασίες μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Επίτροπε. 11 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, έξυπνοι άνθρωποι είστε, δείτε το ρολόι και παρακαλώ να είστε σύντομα. Σύντομοι, με συγχωρείτε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η κυρία Τελκαστία. Είμαι η πρώτη λοιπόν που θα χρειαστεί να αποδείξω την ευφία μου, να δούμε το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο και θεωρώ ότι οι δεσμεύσει της αναφορικά με την καταρχική ημερομηνία προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή κάποιες προτάσεις ε, τηρήθηκαν. Να τις συγχαρώ λοιπόν διότι τίμησε τον λόγο της ε, και τις δεσμεύσεις της. Ε, ακούστηκαν διάφορα μέτρα, αριθμιστικά και άλλα όχι. Μερικά ε, σε αυτόν, ε, όπως η πολιτική του ραδιοφάσματος, είναι ζήτημα πολύ σημαντικό. Και εμείς έχουμε ολοκληρώσει ως Επιτροπή το έργο μας και θα ψηφίσουμε αύριο. Θα ήθελα να προσθέσω λοιπόν στα ζητήματα που ανέφερε η Επίτροπος τα Από θεματικής ένα από τα ζητήματα που αυτή τη στιγμή αποκτούν ένα και πιο σημαντικό ρόλο στην συζητήση μας είναι το cloud computer, το υπολογιστικό νέφος. Το νέφος αυτό όλο και συζητείται στο πλαίσιο της ε, ασφάλειας. Ε, είναι ένα ζήτημα λοιπόν που θα μας απασχολήσει και τους προσεχιούς του προσεχεί μήνε, ε, αλλά και το προσεχέ έτος. Θεωρώ λοιπόν πως ο διατλαντικό διάλογος και η συνεργασία με τι ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Εξάλλου θα ήθελα να τονίσω μέσα σε αυτό το ζήτημα το θέμα των smart grids των εφιών δικτύων που είναι ένα οριζόντιο ζήτημα που αφορά τομείς όπως η ενέργεια για το δίκτυα διανομής αλλά έχει σχέση επίσης και με την ανάπτυξη του διαδικτύου των αντικειμένων των πραγμάτων. Είναι κάτι το οποίο θα αποδά όλο και μεγαλύτερη σημασία στην όλη συζήτηση αλλά και στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν. Και τέλος επιθυμώ να υπογραμμίσω την κεντρική σημασία που είχε, έχει και θα έχει η ψηφιακή ευρωπαϊκή αγορά. Ε, τρόπος αναφέρθηκε σε κάποιες πτυχές όπως η ηλεκτρονική υπογραφή κλπ. Αυτό λοιπόν θα είναι μια σταθερά που θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την Επίτροπο αλλά από, το, ε, από την Επίτροπο και την ιστορική αγορά και θα πρέπει να αποφερθούμε από όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η, κοινωνία, η ψηφιακή κοινωνία. Υπάρχουν δύο θέματα. Το εθίξατε πρόκειται για την διάσκεψη που θα διεξαχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και το φόρουμ για την διακυβέρνηση του διαδικτύου που έχει και αυτό την σημασία του, τη μεγάλη σημασία του μάλιστα. Και πάνω στο ζήτημα αυτό γίνονται πολλές συζητήσει ε, και εργασίες. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσετε και λίγο χρόνο σε αυτό. Αυτά. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την επίσκεψή σας και για τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας και για την γενική παρουσίαση των θεμάτων του χαρτοφυλακίου σας. Είμαστε όλοι εντυπωσιασμένοι για το τι θα κάνετε τους επόμενους μήνες και βλέπω πως ε, θα μπείτε ενεργά στην, στις διαβουλεύσεις. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα συγκεκριμένα σε δύο-τρία θέματα. Είπατε πως ε, θα παρακολουθήσετε την εφαρμογή του τηλεπικοινωνιακού πακέτου και θέλω να σας ρωτήσω ανοιχτά. Εμείς συμφωνούμε όλοι πως το γρήγορο διαδίκτυο για όλους στην Ευρώπη είναι το α και το ω για να υπάρχει ο ψηφιακός κόσμος στο σπίτι. Είστε ικανοποιημένοι με την πρωτοβουλία περί ευρυζωνικότητας. Ε, ε, υπάρχουν αρκετές ε, ιδιωτικές επενδύσεις, υπάρχουν κίνητρα. Είπατε πως είσαι επαφή και με την ΠΕΡΕΚ. Τι σας λένε, δηλαδή από τη Γερμανία μπορώ να σας πω πως ασχολούμαστε εδώ και χρόνια, αλλά έχω την αίσθηση πως δεν προχωράνε αρκετά γρήγορα τα πράγματα και αν είναι να είμαστε και διεθνώς ανταγωνιστικοί είναι όπως είπα η αρχή και το τέλος η ευρυζωνικότητα. Τι θα κάνετε λοιπόν για να συμπληρώσετε αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει. Δεύτερον, αφορά την εξέλιξη του διαδικτύου, έχουμε αναφερθεί σε διάφορα θέματα κατά καιρού. Εσείς αναφέρατε την ουδετερότητα του δικτύου και το τι θα γίνει σχετικά. Ξέρετε πως εμείς κάναμε μία δημόσια διαβούλευση πέρσι και καταλήξαμε πως ε, δεν ξέρουμε αν χρειάζεται κάποια σχετική ε, ρύθμιση ή μήπως βλέπετε ε, εσείς ε, κάποια τέτοια ανάγκη. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω τι άποψη Για την περιαγωγή στα κινητά έχουμε τον δεύτερο κανονισμό περί περιαγωγής ε, και έμαθα πως είπατε σε μια διάσκεψη πως έχετε στόχο μέχρι το 2015 οι διαφορές να μειωθούν μεταξύ, δηλαδή οι διαφορές τιμών εθνικών και περιαγωγής και το ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει εδώ πέρα. Υπάρχει ίσως μια πρόταση για ένα κανονισμό ε, roaming 3. Σε ποια κατεύθυνση θα πάει. Εάν προγραμματίζεται κάτι για μετά τις 26 του 2012 θα σας ευχαριστούσα να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Τέλος, για το σύννεφο των υπολογιστών. Οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Ελευθεριών βεβαίως είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με το θέμα. Θα ήθελα να βερθώ σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Ντελκαστήγιο γιατί ξέρετε πως οι συνάδελφοί μας πάνε στην Ουάσιγκτον για τον υπερατλαντικό διάλογο που θα αφορά και τα προσωπικά δεδομένα και τις συμφωνίες που υπάρχουν με τους Αμερικανούς. Ε μπορείτε να μας πείτε λοιπόν κάποια πράγματα εδώ πέρα για την στρατηγική σας, ευχαριστούσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και αναμένω τον διάλογο μαζί σας ο κύριος Φανίστελ και να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε λίγο στα δύο λεπτά. Ε, σας ευχαριστώ. Θα, θα προσπαθήσω. Δύο ε, θέματα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την παρουσίαση ε, του προγράμματός σας που είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα τον ε, Γαλιλαίο. Ξέρετε πως στην Επιτροπή μας στηρίζουμε το πρόγραμμα αυτό για τις μελλοντικέ ιδιαίτερα προοπτικές που έχει όσον αφορά την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά μας στον κόσμο. Το ζήτημα είναι πως οι υπουργοί δεν ε, μπόρεσαν να βρουν μια μια λύση εντός του προπολογισμού. Δεύτερον, να αφαιρθώ και εγώ στην περιαγωγή, εάν δείτε τα εθνικά νούμερα, Βλέπετε πως μετά το ε, όριο που ετέθη το 2007 μειώθηκε πάρα πολύ το, το κόστος και έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα ε, για το στόχο που έχετε το 2015 να είναι ίδιες οι τιμές οι εθνικές και ε, της περιαγωγής. Ε, ερωτώ λοιπόν, θα θέσετε ξανά ε, ανώτατο όριο. Γιατί λέτε και μάλλον λένε πως αυτό είναι κατά των κερδών επιχειρήσεων. Μπορεί να έχει και κέρδη και με ε, ένα πλαφόν. Η κυρία Τίκαου. Είμαι η πρώτη ομιλήτρια μετά από τη όλε τι που λαμβάνει το λόγο και θα ήθελα να επωφεληθώ τη ευκαιρία προκειμένου να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο και να την ε, ευχαριστήσω για την παρουσία της. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με την χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά το το εμπιζωνικό δίκτυο. Θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι οικονομικοί πόροι, ποιο είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο έχετε προβλέψει και τι μέτρα επίσης προβλέπετε για το θέμα της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του διαδικτύου. Επίσης να αναφερθώ και στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Νομίζω ότι εδώ δεν έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδος, μόλον ότι έχει γίνει αρκετή πρόοδος και σκέφτομαι τα προγράμματα τα οποία εγκρίθηκαν το 2001 και τα οποία ξεκίνησαν να εφαρμόζονται σε κάποια κράτη-μέλη. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες ε, για την περαιτέρω πρόοδησή τους και υπήρχε μια ρύθμιση προκειμένου το 50% των ε, δημοσίων προμηθειών να υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου, άρα απέχουμε πολύ από αυτό το όριο το 50% που είχε τεθεί. Επίσης ε, το ζήτημα της ηλεκτρονικής ε, υπογραφής έχει ιδιαίτερη σημασία να προωθηθεί περαιτέρω. για την αμοιβαία αναγνώριση τώρα αυτών των ε, ηλεκτρονικών υπογραφών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το απαραίτητο για να μπορέσουμε να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση στον τομέα αυτών. Διερωτώμε λοιπόν πότε θα υποβάλλετε όλα αυτά τα όλες αυτές τις προτάσεις γιατί πρέπει να διοργανώσουμε κάποιες ε, συναντήσεις, κάποιες διασκέψεις. Ε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο cloud computing, το υπολογιστικό νέφος, αλλά θα θέλαμε από πλευρά Κομισιόν να δείξετε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση. Ευχαριστώ. Κυρία Ριέρα Μαδουρέλ. Muchas gracias, señor presidente. Ευχαριστώ κύριε Κρούς, εξ ονομέρους της ομάδας μου να σας καλωσορίσω εκ νέου στην Επιτροπή μας και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εργασίες σας και στην εκπλήρωση των στόχων σας και των δεσμευσεών σας. Θα ήθελα σήμερα να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες που καταβάλατε, όπως είπατε, εσείς όλες οι γυναίκες να καταστούν ψηφιακές. Let's get every woman digital. Είναι μια φράση την οποία συμμερίζομαι απόλυτα κυρία Επίτροπε, διότι μόνο 20% των ε, φοιτητών στην ε, δομέα τη μηχανική ή τη πληροφορική είναι γυναίκε, ε, μόνο ότι εκπροσωπούμε πάνω από 50% του φοιτητικού κόσμου ή όπω συμβαίνει στις, με τι γυναίκε, έχουμε ένα χαμηλό ποσοστό ε, ε, διοικητικών στελεχών κλπ. Επίσης ε, θα ήθελα να φροντίσετε προκειμένου να ζητήσετε από τους συνεργάτες σας να ελέγξουν το πώς έχουν οι 101 προτάσεις για που έχουν γίνει αναφορικά με την ισότητα ευκαιριών κλπ. Είπατε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια και τα ερωτήσει που έθεσαν ε, συνάδελφοι να επικεντρωθώ σε μία και μοναδική ερώτηση αναφορικά με την έρευνα και την κοινοτομία. Κυρία Βίτροπε, το ίδιο δηλώσατε εξάλλου, η Κομισιόν θα πρέπει να παρουσιάσει την νομοθετική της πρόταση σχετικά με το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο πριν από τα τέλη ενεστώτος έτους. Όπως και στα προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο, ε, ICTs, το, θα είναι αναφίβολα ένας από τους βασικούς πυλώνες του νέου προγράμματος πλαισίου. Ακούσαμε την πρόταση του συναδέλφου, κυρία Κουίν, για την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία. Ένα, ένα κοινό πλαίσιο λοιπόν, ένα κοινό πλαίσιο για την ε, αγορά και την ε, γνώση. Θα ήθελα να μάθω εσείς ποιο τομέα τονίσατε την στήριξη των ε, αγορών ε, ICT ή στην ε, θέμα των ικανοτήτων και των γνώσεων. Πού βρίσκεται κατά άποψή σας το μέλλον των ICT στα ε, πανεπιστήμια ή στις μεγάλες ερευνητικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Θα ήθελα να μάθω την άποψή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστούμε για την διεξοδική παρουσίαση του προγράμματός σας. Απηχώντας την προηγούμενη ερώτηση για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, θα ήθελα να ρωτήσω Ε, κάτι που σχετίζεται με τα μελλοντικά προγράμματα έρευνας και κοινοτομίας και το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Εξάλλου έχουμε και την πράσινη βίβλο βάσει της οποίας ξεκίνησαν οι δημόσιες διαβουλεύσεις ε, και οι πρώτες ενδείξεις ε, υποδεικνύουν θα πρέπει να έχουμε λιγότερες θεματικές ονενότητες, απλούστερα προγράμματα και απλούστερο πλαίσιο. Ε, το πρόγραμμα πλαίσιο 8 θα καλύπτει πολλούς και διαφορετικούς ε, τομείς. Ε, ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να μεριμνήσουμε και σε νέους τεχνολογικούς τομείς να γίνεται αντίστοιχη έρευνα. Μας είπατε ότι βρίσκεστε σε πρώιμο στάδιο συζήτησης ε, για την ε, καινοτομία και για τον ανταγωνισμό το ICT. Δηλαδή, θεωρείτε ότι θα αλλάξει κάτι σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για τις ε, τεχνολογίες, πληροφορίες, μιλώντας για την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία. Θα αλλάξει κάτι για αυτές τις νέες τεχνολογίες στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Προβλέπετε κάτι τώρα που προετοιμάζετε αυτό το 8ο πλαίσιο. Σας ευχαριστούμε κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε την Επίτροπο για την σημερινή της παρουσία και για την παρουσίαση της ατζέντα. Ε, μιλώντας για το κυβερνοέγκλημα και για την κυβερνοασφάλεια, θα ήθελα να ρωτήσω αν κατάλαβα καλά ότι συγκροτείται ένα νέο σώμα που θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, μια που η παρουσία της είναι πρόσφατη στην Ενίζα, γιατί αυτό το έργο δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε να το αναλάβει η Ενίζα στα γρήγορα. Υποτίθεται ότι αυτός είναι και ο σκοπός της και να μια ευκαιρία, μια που έχουμε και το κυβερνοέγκλημα και την ανάγκη για κυβερνοασφάλεια, να ενισχύσουμε ένα ήδη ιδρυμένο agency της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Ευχαριστώ κύριος De Angelis. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για την ε, παρουσίασή της ε, θα, ε, και έρχομαι στην ε, συζήτηση. Η πρώτη ερώτησή μου ήδη τέθη από τον κύριο Βανίστερο και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη ε, για τον Γαλιλαίο λοιπά. Δεν επανέρχομαι. Τώρα, δεύτερη ερώτηση. Όπως γνωρίζετε, η σύσταση σχετικά με την πρόσβαση στα νέα δίκτυα με οπτικής ίνας είχαν ως στόχο να εγγυηθούν την ανταγωνιστικότητα των νέων δικτύων Τώρα, τα εθνιστικά πλαίσια ορισμένων κρατών, κανένα άποψή μου φαίνεται όπως διαφοροποιούνται από αυτή τη σύσταση. Οι προσεγγίσεις που γίνονται από τα κράτη-μέλη θέτουν σε κίνδυνο την εναρμόνιση των κανόνων και σε ό,τι φορά την συνεκτικότητα, θα πω ότι και η σύσταση αναφορικά με τα τιμολόγια το 2009 θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε μια μείωση των τιμών των κινητών, της κινητής τηλεφωνίας. Σήμερα τέσσερις φορές επί 27 εφάρμοσαν αυτήν την σύσταση του 2009 και όλα αυτά καθυστέρησε τα ωφέλη ειδικά για τους πολίτες, για τους Συνδρομητέ, διατηρώντας την ανισορροπία ανάμεσα στις ε, ε, την κινητή τηλεφωνία και τη σταθερή τηλεφωνία. Σα ρωτώ λοιπόν, Πρόεδρε, ε, ε Επίτροπε, συγγνώμη, θεωρείτε ότι οι ελλείψεις που έχουν παρουσιαστεί σε αυτόν τον τομέα δεν κινδυνεύουν να δημιουργήσουν νέε τρευλώσει του ανταγωνισμού και εν ώψη της ε, μετάβασης στην οπτική ίνα. Και εσείς ε, πώς προτίθεστε να, τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να ολοκληρωθεί η ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Παρακολουθώ εκ του ε, και με απασχολεί ιδιαίτερα, αλλά θεωρώ ότι παράλληλα είναι και ένα εξαιρετό ζήτημα, το Innovation Partnership ε, κλπ. Και εγώ, επειδή είμαι άμεσα ενδιαφερόμενη και έχω μια σύγκρουση συμφερόντων εδώ, διότι λόγω ηλικίας με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, θεωρώ ότι πολλά ότι μιλάμε πάρα πολύ για τα τεχνολογικά ζητήματα, αλλά ελάχιστα για το πώς ε, θα χρησιμεύσει στον χρήστη, στον συνδρομητή. Μιλούσα σε ένα, ένα νοσοκομείο το οποίο ναι, το οποίο θα, θα ήθελε να διοργανώσει ένα μάστερ για νοσηλεύτριες, ε, για το νοσηλευτικό προσωπικό. Και θα ήθελε λοιπόν να μπορέσει να προωθήσει ένα, έναν τρόπο ε, θεραπείας ε, των των ασθενών. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο διαδίκτυο, κάποια ιστοσελίδα, για να μπορέσουμε λοιπόν να γνωρίσουμε και να ενημερωθούμε. Η κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας βλέπω. Είστε μία από τις πιο δραστήριες επιτρόπους και αποδεικνύεται πως οι γυναίκες το κατέχουν το ψηφιακό. Έχω πολλές ερωτήσεις. Συμφωνούμε νομίζω πως η Ουγγρική Προεδρία έχει, ε, τα έχει πάει καλά στην ψηφιακή ατζέντα και Είχαμε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη για τις γυναίκες και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το υπολογιστικό αυτό νέφος. Όταν μιλάμε για την Ευρώπη, μιλάμε πάντα για την ομοθεσία και το περιεχόμενο, αλλά δεν συζητάμε τις απαραίτητες υποδομές. Τι άποψη έχετε λοιπόν για τις στρατηγικές υποδομές που είναι απαραίτητες στην Ευρώπη για Ευρωπαίους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς πρέπει να εξελιχθεί για το μέλλον. Και η άλλη μου ερώτηση, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο, την ανάπτυξη της ε, ψηφιακής ε, ατζέντα. δηλαδή το η δορυφορική ευρυζωνικότητα για την Ήπεθρο και μια που μιλάμε για ευρυζωνικότητα για όλους, μιλάμε για ευάλωτες ομάδες, γυναίκες, ηλικιωμένους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς το βλέπετε αυτό το ζήτημα. Και τέλος πρέπει να σας ρωτήσω. Ξέρετε πως υπέστη επίθεση η σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα πράγματα. Πώς το βλέπετε αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Καλβίνη. Uh, Ευχαριστώ. Επίτροπε, αναφερθήκατε στην εκπόνηση της στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια στο πρόγραμμά σας. Ξέρετε όμως, δεν μπορώ να είμαι τόσο αισιόδοξη. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα τίνω να γίνω άπεσιόδοξος, διότι κανείς δεν θέλει να αναλάβει τα ενία για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα στην Ένωση. Δεν πρόκειται μόνο για την ομάδα ΣΕΡΤ, ε, την ομάδα με σου Υπάρχουν εκατοντάδες ε, παραδείγματα κυβερνοεπιθέσεων, γιατί η κυβερνοεγκληματικότητα δεν περιορίζεται στο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Ε, αναφερθήκατε λοιπόν στην εκπόνηση στρατηγικής για το θέμα αυτό και το επιδοκιμάζω. Ποιος όμω θα τεθεί επικεφαλής ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς? Ε, γνωρίζω ότι τίθενται και θεσμικά ζητήματα. Ε, χρειάζεται συντονισμό λοιπόν όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια. Δεν θα ενεργήσετε μόνοι σα. Για το υπολογιστικό νέφος τώρα. Ε, φυσικά θέλουμε να συμμετάσχουμε στις διαβουλεύσεις και θέλουμε μέχρι το 2020 να έχουμε μια στρατηγική για το cloud computing, γνωρίζοντας ότι θα επέλθουν αλλαγές στην νομοθεσία μετά τη θέση σε λειτουργία της ε, στρατηγικής, μετά τη θέση εφαρμογή κάποιων ε, νομικών πράξεων. Πώς σκοπεύει να κινηθεί τα επόμενα τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω να είστε έτοιμοι πριν περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια. Είναι μακρύς ο δρόμος και πώς ε, ε, προτίθεστε εσείς να προετοιμαστείτε πριν ε, αρχίσετε να τον ακολουθείτε. Ο κύριο Φέκμαρκ, ευχαριστώ, θα είμαι σύντομο. Δεν ξέρω αν η κυρία Επίτροπο θα ήθελε να μας πει το πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει την ταχύτητα των εξελίξεων παγκοσμίω τι κάνουμε όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά μας σε σχέση με την πραγματική ανάπτυξη και τις εξελίξεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Απλή ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο για να απαντήσει στις πολλές και διαφορετικές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση του κυρίου Χέκμακ μοιάζει ευκολότερη αλλά είναι πιο δύσκολη. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε πάντα, έτσι να το πω κάπως διπλωματικά, ε, δεν μπορούμε πάντα να πούμε ότι θα το κάνουμε εμείς ό,τι θέμε, χαλαρά κτλ. Ε, γιατί δεν είμαστε ε, έτσι, τόσο άνετοι από πλευρά χρόνου. Αυτό φαντάζομαι εννοεί ο κ. Χέκμαρκ. Γνωρίζουμε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, εξελίξεις δηλαδή από Ανατολή είναι πιο δραστήρια όχι μόνο όσον αφορά την παραγωγή όλων αυτών των πραγμάτων που χρειάζονται αλλά έχουν και τα ακαδημαϊκά, αυτά, τα ακαδημαϊκά προγράμματα για την παραγωγή αυτών των μηχανικών που χρειάζονται για τους υπολογιστές. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο αποφύτους στο έτος. Ακόμα και αν δεν δραστηριοποιηθούν όλοι αυτοί σε αυτόν τον τομέα, ε, σας διαβεβαιώ πως όταν έχουμε τέτοια νούμερα και αν τα συγκρίνουμε με την, με την Ευρώπη, η Ευρώπη είναι σταγόνα στον ωκεανό. Βλέπουμε πως ε, πλέον δεν μιλάμε μόνο για ένα μεγάλο ανταγωνιστή, αλλά ε, βγάζουν και τους ανθρώπους αυτούς που θα κάνουν αυτές τις εξελίξεις. Λαμβάνοντας λέει υπόψη πως ε, στη Silicon Valley η παραγωγή περιεχομένου είναι εντυπωσιακή ακριβώς όταν συζητάμε ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης νομίζω πως δεν έχουμε χρόνο να είμαστε χάλαροι για να αναπτύξουμε μια στρατηγική ε, και να καταλήξουμε σε μια συνένεση. Πρέπει να ξέρουμε και βεβαίως το αξίζουμε και πρέπει να το κάνουμε πως πρέπει να επιταχύνουμε. επίσης μιλώντας για το ζήτημα των γυναικών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά γενικότερα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τόσους πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους. Αλλά όταν ξεκινάει κανείς ε, καθυστερημένα και δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, τότε δεν μπορεί κανείς να ε, αναπληρώσει αυτό το, το κομμάτι και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε η κυρία Μαντουρέλ και Χέρτσοκ. Και άρα η πρωτοβουλία αυτή που έλαβαν κάποιες γυναίκες από τον κόσμο της πληροφορικής να κάνουν προγράμματα για κορίτσια 10 ετών. Έτσι, πληροφορίες. Και το υπόβαθρο που χρειάζονται, το τεχνικό, το μαθηματικό και το τα λοιπά, όπου κατά κανόνα τα κορίτσια λένε ότι δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Προσπαθούν λοιπόν να τους κάνουν να ενδιαφερθούν, να τους πούν ότι είναι συναρπαστικά, είναι τόσο κοντά στην κοινωνία. Αλλά ε, όπως είπα πρέπει να ξεκινήσουμε με τα κορίτσια των 10 ετών, όταν ακόμα το μυαλό τους είναι ανοιχτό και μπορούν να επιλέξουν το ποια εκπαίδευση θα ακολουθήσουν. Free every Πρέπει λοιπόν να του λάβουμε όλους υπόψη για ε, να δούμε τι θα κάνει η Ευρώπη στον τομέα αυτόν. Και αυτή είναι η πρόκληση εδώ πέρα αυτού του χαρτοφυλακίου, γιατί το χαρτοφυλάκιο είναι οριζόντιο, είπαμε συνδέεται με όλους αυτούς τους τομείς και με τον Τζον Ντάιλι και με την Σεσίλια Μάρμστλο μιλήσαμε για την ε, κυβερνοασφάλεια και μια που λέμε για το ότι πρέπει να γίνει ψηφιακό ο κάθε Ευρωπαίος ε, να μην είναι ξένη γλώσσα αυτά τα πράγματα αλλά εάν πούμε κάτι τέτοιο ε, θα μου πούν οι Ευρωπαίοι μπορείτε να μας δώσετε ασφάλεια αλλιώς αφήστε δεν πειράζει δεν με ενδιαφέρει αν είναι να μην έχω ασφάλεια και ακριβώς εδώ πέρα η Σεσίλια Μάλστρομ που βεβαίως ε, έχει την κυβερνοεγκληματικότητα και εγώ για την κυβερνοασφάλεια συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να ασχοληθούμε με αυτό το ε, ζήτημα. Και βέβαια θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τους υπουργούς στην Ουγγαρία και μέρος ε, βεβαίως θα το παρακολουθήσει και ο Αμερικανός συναδελφός μας, ο αρμόδιος για την εσωτερική ασφάλεια και νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε ούτως ή άλλως ε, το πάνε για να δοθεί έτσι περισσότερη ουσία σε αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ασφάλεια 100% όχι. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Η ζωή, ξέρετε, ορισμού τα φέρνει έτσι. Αλλά Πρέπει να το, να το δούμε αυτό το ζήτημα. Είχατε και την εμπειρία της προηγούμενης εβδομάδας και η Κομισιόν πριν από λίγες εβδομάδες, της επίθεσης δηλαδή, οπότε δεν είναι κάτι μακρινό. Είμαστε και ενδιαφέρον στόχος και πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πιο ασφαλή. Πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και ο Μάρος Σεύκοβιτς και εγώ καταφέραμε να συναντηθούμε και ευχαριστώ εδώ πέρα και το Κοινοβούλιο και να συνεργαστούμε γιατί το Κοινοβούλιο ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό και βρήκαμε μια γραμμή έτσι για να συνδέσουμε όλες αυτές τις διάφορες μονάδες που εμπλέκονται και να μην μιλάμε για φέουδα του καθενός εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Hackers, to say, Όσον αφορά τώρα την Ενίσα, παίζει ρόλο κλειδί σε αυτό και στηρίζει με την πείρα της ε, αυτές τις δραστηριότητες. Και πράγματι θα πρέπει να καλύψουμε την Ευρώπη ε, εντάξει, κάποια τα πάνε ήδη πολύ καλά, κάποια είναι λίγο ε, πίσω, αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την, την εμπειρία που υπάρχει και της ε, ΕΝΙΣΑ και των κρατών μελών που είναι μπροστά η ομάδα εργασία με τι ΗΠΑ για την ε, κυβερνοεγκληματικότητα τα πάει καλά υπό την ηγεσία της ε, Σεσίλια και το παρακολουθούμε κι εμείς. Οπότε νομίζω πως ε, δεν πρέπει να σπαταλάμε χρόνο συζητώντας περί αρμοδιοτήτων και εγωισμών. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για τον Γαλιλαίο και το πόσο ενδιαφέρον είναι. Όσο ενδιαφέρον και αν είναι δεν είναι δικό μου θέμα και ο Αντώνιο ο συνάδελφος είναι υπεύθυνο, αλλά εάν μου επιτρέπετε να κάνω μια προσωπική παρατήρηση αυτές οι νέες αντιπαραθέσεις με τον προϋπολογισμό και τον νέο προϋπολογισμό και τους νέους προϋπολογισμούς ε, δεν είναι σωστές. Πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση αυτών των έργων και όχι μόνο έτσι να βλέπουμε την τεχνική σκοπιά, του, του Για να επανέλθω στα της αρμόδιότητάς μου, η έρευνα που ανέφεραν αρκετοί από σας Είχαμε εκεί πέρα καλή συνεργασία με τη Μόρα. Κάνει καλή δουλειά. Και μην με παρεξηγείτε. Ε, όλοι οι συνάδελφοι είναι καλοί. Εξορισμού είναι όλοι καλοί. Ε, καμιά φορά τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά έχουμε την ίδια προσέγγιση όταν μιλάμε για την έρευνα και τι συνάδελφος συμφωνεί απολύτως για το ότι θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση για τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και για το ότι και η βασική έρευνα ε, στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική για να ανθίσουν έτσι πολλές πρωτοβουλίες. Έγινε μια ερώτηση για το εάν είναι συναρπαστικό να βγει κανείς εκτός του εργαστηρίου και για την καινοτομία του προγράμματος πλαισίου 8. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το πρωί για μια αντιπροσωπεία και το τι διακυβεύεται. Και τα ερευνητικά ιδρύματα και η βιομηχανία και όσοι τελικά εμπλέκονται μετά την εφαρμογή όλοι να λένε παρακαλώ εκμεταλλευτείτε, σας παρακαλούμε εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία του προγράμματος πλαισίου 8 και βεβαίως αυτό σχετίζεται με τη στρατηγική του Γκέναρ για το τι διακυβεύεται στην Ευρώπη και πώς πάλι το πώς πάλι θα έχουμε την καινοτομία σε πρώτο ρόλο Έχουμε εξαιρετικούς ερευνητές, έχουμε καινοτομία και εξαιρετικές προτάσεις, οπότε δεν είναι θέμα ε, του ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ευρώπη. Είπα, έχουμε εξαιρετικά ερευνητικά Ινστιτούτα και παράγεται καινοτομία. κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να είστε περήφανος για κάποια από αυτά που βρίσκονται στη χώρα σας, αλλά αυτό είναι σύμπτωση, θα έλεγα, γιατί είναι ευρωπαϊκή η προσπάθεια. Και ξέρετε πως ε, σημαντικό είναι να συνδυάζουμε τις προτάσεις μας. Τώρα, το υπολογιστικό νέφος είναι συναρπαστικό και ε, οπωσδήποτε πρέπει να το συζητήσουμε ε, εξετάζοντας το μέλλον της Ευρώπης. Οπωσδήποτε πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω την πολιτική μας ε, και το ταχύτερο δυνατόν μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό και δεν θα πρέπει ε, να ακολουθήσουμε τη γραμμή ε, της αναμονής, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα προλάβουμε. Οι επενδύσεις στο υπολογιστικό να έχουν στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, γιατί μόνο έτσι θα γίνει πραγματικό αγαθό ο υπολογιστής για όλους. Και σε αυτό αποσκοπούμε, γι' αυτό προσευχόμεθα και αγωνιζόμεθα. Έξωθεν ε, ε, έρχονται διάφορες ε, πρωτοβουλίες και πρέπει να ακολουθήσουμε. Χρειαζόμαστε ριζοσπαστική δράση για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γι' αυτό εξήγηλα διαβούλευση τις ερχόμενες εβδομάδες και σας διαβεβαιώ ότι συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για μας το θέμα αυτό. Το θέμα, το βασικότερο θέμα είναι το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής. Ε, θα είναι πραγματικά συναρπαστικό το θέμα, αλλά σας λέω δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να ε, ρυθμιστούν και να λυθούν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Για την περιαγωγή τώρα, οι τωρινοί κανόνες ε, περί έχουν ε, προς το παρόν προστατεύσει τους καταναλωτές ενάντια στις υπερβολικές τιμές, αλλά τώρα μιλάμε για την επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός, δεν υπάρχει σωστή δυναμική στις τιμές της λιανικής ε, για, τα, για την μεταφορά δεδομένων ε, και για την περιαγωγή γενικά. Άρα θα πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο και προτείνω μια υβριδική προσέγγιση. Φαίνεται λίγο, ακούμε σαν θαυματουργός, αλλά αυτό χρειάζεται. γιατί έτσι θα υπάρχουν σταθερές και πάγιες υπηρεσίες περιαγωγής στο μέλλον για τους καταναλωτές και θα καλυφθεί το, σε χαμηλότερες τιμές ε, και θα καλυφθεί το θέμα της ε, προστασίας και της ασφάλειας. θα ήθελα να σας δώσω και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Ε, το Μάρτιο ε, οι διευθύνοντες ε, σύμβουλοι μεγάλων ε, τηλεπικοινωνιακών εταιριών με προσκάλεσαν σε διάλογο παρευρέθηκαν και διάφοροι άλλοι φορείς του ιδιωτικού τομέα, επίσης μεγάλες ραδιοτηλεοπτικές εταιρείε. Ακόμη και ο Steve Jobs ήταν μαζί μας online βέβαια γιατί δεν μπορούσε να έρθει για λόγους υγείας. Δεν συμφώνησε ο γιατρός του να ε, κάνει το αεροπορικό ταξίδι. Επίσης είχαμε τους ε, κατασκευαστές που εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση. Σε αυτή την ευρεία διάσκεψη συμφώνησαν όλοι ότι χρειαζόμαστε ρηξικέλευθο τρόπο σκέψης και πρέπει ε, με τις πράξεις μας να δείξουμε ότι είμαστε όντως δημιουργικοί. Εάν στον τομέα σας, αν στη χώρα σας μπορέσετε εσείς να αποδείξετε ότι είστε αρκετά ικανοί και μπορείτε να το κάνετε, τότε ε, δεν θα έχω προφανέστατα κανένα πρόβλημα γιατί εσείς θα διαχειριστείτε ε, το έργο σας, θα υπομιστείτε την ευθύνη σας για τη δραστηριότητα που έχετε αναλάβει. Τι συζητείτε τώρα, τι διακυβεύετε. Ή μάλλον να σας πω ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τέσσερις ομάδες εργασίας ε, Ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Deutsche Telekom ηγείται, προεδρεύει μόνο σε μία μοδέα. Ο κύριο Λέβη τη Βιβέντη προεδρεύει τη δεύτερη. Ο Μπεν Φορβάε, μια ε, εκπρόσωπο κατασκευαστική εταιρεία που στο, στην τρίτη ομάδα εργασία, όλοι μου υποσχέθηκαν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στην προβλεπόμενη προθεσμία ε, ε, για να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις δημιουργικές και ενωτόμες, ούτως ώστε να αλλάξει άρδιν το σκηνικό. Εάν αυτό δεν αποδειχθεί αληθινό ε, αν δεν αν ε, δεν μας δώσουν τα υπεσχημένα, τότε θα αναλάβω εγώ ηγετικό ρόλο. Πάντως, η στρατηγική της Ευρώπης στον τομέα έχει τέτοια βαρύτητα που θα πρέπει να τους εγκαλέσουμε όλους να επομιστούν τις ευθύνες τους εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων. Αλλιώς θα αναλάβουμε διαφορετική δράση. Για την ηλεκτρονική υπογραφή τώρα, και τις σχετικές ευρωπαϊκές αποφάσεις ε, ε, κατέγραψα το περιεχόμενο των ψηφισμάτων. Τώρα για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών ε, διεπαφών, κυρίως όταν μιλάμε για την διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών. Ε, όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και θα επανέλθω. Εντάσσεται όμως το συνολικό πακέτο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οπότε έχουμε αναλάβει συγκεκριμένη δέσμευση στην υπηρεσία μου και εγώ προσωπικά να κάνουμε τις απαιτούμενες προσπάθειες ε, ούτως ώστε να υπάρχει αναγνωρισιμότητα, να λειτουργήσει το σύστημα των υπογραφών μέσα στην ενιαία αγορά. Είπα στον συνάδελφό μου τον κύριο ε, Μπαρνιέ ότι εγώ με το μέρος σου είμαι, αλλά είναι αμφίδρομη η συνεργασία. Δηλαδή κάτι θα πρέπει να δώσετε κι εσείς για το θέμα των πνευματικών ε, δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε το ένα θέμα χωρίς το άλλο, αλλιώς πάρτι με ένα άτομο δεν γίνεται. Κίνητρα υπάρχουν. Γνωρίζετε την Επιτροπή Κώστην Ευρωπιάνα Και θα αντιλαμβάνεστε κι εσεί ότι αν δεν λύσουμε το πραγματικό πρόβλημα των ορφανών έργων, ε, παραδείγματο χάρη, ή γενικότερα των ε, δικαιωμάτων επνευματική ε, ιδιοκτησία και μιλάμε μόνο για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, θα είναι η μη τελή η λύση που θα δώσουμε. Χρειαζόμαστε σφαιρική λύση. σχετικά με την εφαρμογή των αθεωρημένων πακέτου τηλεπικοινωνιών, όπω σα έλεγα, δεν θα διστάσω. Θα εκκινήσω διαδικασίε σε παραβάσει αν κρίνω ότι είναι αιτιολογημένε. δεν ναι, φοβούμε να αναλάβω τέτοιου είδους δράση. Ένα λεπτάκι, ξέχασα κάτι για την περιαγωγή πάλι. Όχι, το ολοκλήρωσα, το ίδιο και το υπολογιστικό νέφος. Σας μίλησα για τη 13η Ιουλίου. εδώ. τελείωσα. Sehr Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές και τον χρόνο που αφιερώσατε. Οπότε τελειώσαμε και με αυτό το θέμα της μερικής διάταξης. Οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε τους μήνες που έρχονται και περνάμε στο επόμενο σημείο. Δηλαδή, εξέταση του εβδομού προγράμματος ε, πλαίσιο υπαρχμών 7. Und ich darf... Ε, πρώτα απ' όλα να δώσω τον λόγο στον κύριο Οντί, τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στο πλαίσιο της ε, συζήτησης των τροπολογιών και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Στον χρονοδιάγραμμα υπενθυμίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε με μεγάλη καθυστέρηση ανακοίνωσή του το Φεβρουάριο 2011 και πως ε, για να μπορέσει να εκφραστεί το Κοινοβούλιο κάτω από συνθήκες που θα είναι χρήσιμες αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε ένα χρονοδιάγραμμα πολύ πιεσμένο. Θα ήθελα να ευχαριστώ τη Γραμματεία, τον κύριο Γκέο και τη Σουζάν Κίφερ αλλά και τους πολιτικούς συμβούλους, Αλφέντο Σούζα, Ελιζαμπέτα Μοντάνο και τη συνεργάτη μου Φεν Ορλέη. Εντάχει κάποιες πληροφορίες, 308 τροπολογίες ε, κατατέθησαν και προτείναμε σε όλες τις πολιτικές ομάδες ε, διάφορες ε, συμβαστικέ προτάσει ε, αφορούν την ε, θέμα τη εδαφικότητα, ε, τη διαπλούστευση, τη συμμετοχή των γυναικών, την έρευνα, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, την άμυνα και θα επανέλθω εντό λίγου, αλλά και τους στόχους τη στρατηγική 2020. συνεργαστήκα με τους κοιόδες συζητητές. Ευχαριστώ. Μπρίδα Τόμψεν, δεν ξέρω αν παρευρίσκεται. Έλενα Χένκ, Φιλιπ Λάμπερ, Αντιφόρμ, Ζαματίας, Καταρτήσαμε λοιπόν 30 συμβαστικές τροπολογίες, ε, τις οποίες ε, υπέγραψαν τέσσερις πολιτικές ομάδες, τις 17 εξ αυτών και τις υπόλοιπες τρεις πολιτικές ομάδες. Μία μόνο συμβαστική τροπολογία απερίφθη, αυτό που αφορά στην άμυνα. Αναφέρομαι τώρα στις συμβαστικές τροπολογίες, υπάρχουν τέσσερα. Ε, αναφερθήκαμε στην προστέμενη ευρωπαϊκή αξία σχετικά με την αρχική εκδοχή της όπου είχαμε εκφράσει, είχαμε πει μάλλον ότι η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία δεν ήταν προφανής αλλά τελικά το κάναμε πιο θετικό το έγγραφο με πολλές τροπολογίες για την απλοποίηση. Χαιρετίζω τη Μαρία Καβάγιο που έκανε μια εξαιρετική εργασία πάνω στο θέμα. Ε, παραλαμβάνουμε αυτήν την βούλησή μας προκειμένου να πετύχουμε την απλοποίηση συμπεριλαμβανομένων και των ε, καταστάσεων του παρελθόντων. Η τροπολογία 16 αντικαθιστά μια παράγραφο για την εδαφικότητα. Πρόκειται για έναν συμβασμό ο οποίο ε, ήταν δύσκολο να καταρτιστεί για να το συντάξουμε. Θέλαμε να έχουμε καλύτερη συνοχή μεταξύ του έδου προγράμμου πλησίου και των διαθροντικών ταμείων, διότι διατηρώντας την αρχή της αριστείας σε θέματα ευρωπαϊκής έρευνας, να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη, μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των κρατών μελών που μέχρι τώρα δεν συμμετέχουν επαρκώς στο Ταμείο της Έρευνας και να αναπτύξουμε τις ε, σχετικές υποδομές. Ο συμβασμός υπαρθμών 17 αφορά στη συμμετοχή των γυναικών και φτάνω στο πρόβλημα που άπτεται της άμυνας ε, έγραψα ένα, μια παράγραφο μάλλον σχετικά με το θέμα ότι ήγγικεν η ώρα προκειμένου να εξετάσουμε πώς σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έρευνα σε ζητήματα άμυνας. Φαίνεται, σύμφωνα με την άποψη ορισμένων εμπειρογνωμόνων, ότι έχουμε καθυστερήσει διότι η έρευνα σε ζητήματα Άμυνα ε, κοστίζει ιδιαίτερα, είναι πολύ δαπανηρή και υπάρχει σπάνης ε, δημοσίου χρήματος ε, και θα μπορούσαμε λοιπόν να ε, χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τα κονδύλια στον, του τομέα της άμυνας. Κάποιες χώρες το πράττουν σε ενημέρες επίπεδο. Η χώρα στην οποία ανήκω μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζονται και σε το ερώτημα στο Κοινοβούλιο αν δεν θα έφτασε η κατάλληλη στιγμή με την νομική βάση που αναφέρεται στην έκθεση, δηλαδή στηριζόμενη στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, να α, έχουμε μια απαρχή, ένα ταμείο έρευνα ένα ταμείο, όχι ένα ταμείο, αλλά μια πολιτική ε, έρευνα σε θέματα άμυνα που χρηματοδοτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που θα στηρίζει την αμυντική μα βιομηχανία. Ε, υπάρχουν διάφορα κείμενα που προτάθησαν από την κυρία Καστίγιο, την κυρία Μαντουρέλ. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σας για να γνωρίζω κατά πόσο το Κοινοβούλιο μπορεί να εξεύρει μια μια ψηφία έτσι ώστε να αποστείλει ε, σχετικό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Τροπή και τον επιμένω σε αυτό το σημείο ότι έφτασε η ώρα προκειμένου να ε, αποστείλουμε αυτό το μήνυμα με ένα κείμενο το οποίο θα πρέπει να χτενίσουμε μέχρι αύριο και εν ώψη της Ολομέλειας θα μπορούσαμε να βρούμε μια διατύπωση η οποία θα αρμόζει και θα βρίσκει σύμφωνε όλε τι πολιτικέ ομάδε. Αυτά, Πρόεδρε, συνοψίζονται στι 29 ε, συμβαστικέ τροπολογίε που θα ψηφίσει η Επιτροπή μα αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα το λόγο έχει ο κ. Τσουκαλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, λαμβάνω το λόγο για να ευχαριστήσω κυρίως τον συνάδελφο τον κύριο Ντί για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στην έκθεσή του αλλά και την ε, κοπιώδη και αξιόλογη προσπάθεια να συγκεντρώσει τις πολυάριθμες τροπολογίες που προτάθηκαν και να καταρτήσει σοφές συμβιβαστικές προτάσεις. Επί του αντικειμένου, επί της ουσίας, ε, έχουμε ένα πολύ σοβαρό κείμενο για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό το ακούσαμε να στο λέει και η απελθούσα επίτροπος η κυρία Κρούς, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς επίσης και το ζήτημα το οποίο η έκθεση της κυρίας Καρβάλιο αντιμετώπισε, της απλούστευσης, είναι τα δύο ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερο αισιόδοξο για την επίτευξη των στόχων του 2020. Τίποτα δεν μας δείχνει από τα στοιχεία που δημοσιεύονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση που συμβαίνει επειδή η επιστήμη παγκοσμιοποιείται, η έρευνα γίνεται δικτυακή και τα έθνη υποχωρούν μπροστά στις ενώσεις του. Στις 28 Μαρτίου η Royal Society of London δημοσίευσε μία σπουδαία μελέτη την οποία επιγράφει knowledge, networks και nations από την οποία δανείζομαι μερικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 εκατομμύρια ερευνητές στον κόσμο. Η ετήσια δαπάνη για τεχνολογία και ανάπτυξη είναι 1.100 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής, έχοντας σημειώσει 45% αύξηση από το, από το 2002. 25.000 ε, επιστημονικά περιοδικά δημοσιεύουν 1,58 εκατομμύρια άρθρα κάθε χρόνο, εκ των οποίων το 20% ανήκει στην Αμερική, που ξοδεύει και τα 400 δισεκατομμύρια του ετησίου κόστους που σας ανέφερα. Το 35% από τα άρθρα αυτά είναι συνεργατικά. Οι νέες αναδυόμενες χώρες που και πριν αναφέρθηκαν έχουν επιφέρει μείωση των επιδόσεων ε, της Αμερικής για παράδειγμα η οποία από το 1996 έως το 2008 20, έχασε το 20% το 1 πέμπτο δηλαδή από το ποσοστό των δημοσιευμάτων της η Ιαπωνία του 22% και η Ρωσία του 24%. Οι επενδύσεις στην Ευρώπη δεν είναι τόσο υψηλές. Η Κίνα επενδύει με ρυθμό επενδύσεων 20, αύξησης 20% το χρόνο από το 1999 έχει φτάσει στο 1,45% του ΑΕΠ και εξοδεύει 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο στοχεύοντας το 2,5% το 2020. Όσο δε για το πόσους μηχανικούς χρειαζόμαστε ή όχι, ανέφερε η κυρία Κρούζ ένα νούμερο, να αντιπαραθέσω εγώ το 1,5 εκατομμύριο μηχανικούς και επιστήμονες που παρήγαγε η Κίνα το 2007 και τα 2,5 εκατομμύρια που παρήγαγε η Ινδία κατά το ίδιο διάστημα. Επομένως, πρέπει να πάρουμε επίγοντα μέτρα, επίγοντος χαρακτήρα, μια που αν δεν είναι απλώς εμβληματική ορολογία η έρευνα και η καινοτομία αλλά πράγματι η ευρωπαϊκή ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί επάνω σε αυτό ακριβώς τότε είναι προφανές ότι παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες πρέπει να κάνουμε ως προς την απλοποίηση όχι μια εξέλιξη evolution αλλά μια revolution έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι δυνάμεις που σήμερα καταπιέζονται των επιστημόνων από τη γραφειοκρατία για να μπορέσουν να επιδοθούν με μεγαλύτερη άνεση στις έρευνές τους. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που μίλησα πολύ. Η κυρία Ματίας κατόπιν. Και εγώ είχα ζητήσει το λόγο μόνο και μόνο για να ευχαριστήσω και να να τον κύριο Ντί και να τον συγχαρώ για τις προσπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να συμπεριλάβει στο κείμενο του όλες τις ε, θέσεις που εκφράστηκαν κατά το δυνατόν φυσικά. Κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για να λάβει υπόψη τις επιθυμίες μας και τα σχόλιά μας. Και με τις συμβαστικές τροπολογίες ε, θεωρώ ότι κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε μια θέση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για το έργο που θέλουμε να επιτύχουμε. Κρίνω λοιπόν ότι οι συμβασμοί αποτελούν και συνοψίζουν την διαφορετικότητα που υπήρξε και πρόκειψε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Όπως ε, προείπα, δεδομένου του έχω καταθέσει τροπολογίες οι οποίες ε, λήφθησαν υπόψη από τον εισηγητή και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Φυσικά δεν μπορούσα να, να ε, πω ότι έγιναν 100% δεκτές οι τροπολογίες μου, αλλά με στόση η συμπερίληψή τους ε, στις ε, συμβαστικές τροπολογίες ε, με ικανοποιεί. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή για την προσπάθεια τώρα που σε ό,τι φορά την άμυνα δεν είναι τυχαίο πως αυτό είναι ένας τομής επί του οποίου συμφωνούμε αλλά πρόκειται για ένα ζήτημα που συχνά δημιουργεί διεστάμενες απόψεις. Ε, θεωρώ ότι αυτή είναι μια περίπτωση που μας προσφέρεται προκειμένου να ε, προωθήσουμε ένα κείμενο το οποίο θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό με, από τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία των συναδέλφων και να δώσουμε κοινή απάντηση. Η κυρία Εκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Οντί για το εξαιρετικό του έργο και για την διάθεσή του για συνεργασία. Έχω όμως κάποια ερωτηματικά ακόμα και κυρίως θεωρώ πως πρέπει να δούμε το ζήτημα του ότι απομακρύνεται η βιομηχανία από τα ερευνητικά μας έργα. Δεν μιλάμε μόνο για τις μικρόμεσες επιχειρήσεις. Εάν δούμε συνολικά το ποσοστό των προγραμμάτων πλαισίου των τριών τελευταίων, θα δούμε πως η συμμετοχή της βιομηχανίας μειώνεται. Και μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Επίσης, διστάζω λίγο, για τη διατύπωση που έχετε εκεί πέρα για την εδαφική έρευνα. Δεν ξέρω αν είναι γλωσσικό το ζήτημα. Αυτό το οποίο λέτε πως θα πρέπει να υπάρχει ε, ίση χρηματοδότηση μεταξύ των πανεπιστημίων και να, είναι, ε, να έχει εδαφική βάση η έρευνα. Νομίζω πως η αριστεία είναι σημαντική όταν μιλάμε ε, γενικώ για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και εκεί πέρα στοχεύουμε. Και το άλλο ζήτημα στο οποίο έχω κάποιους δισταγμούς αφορά το ζήτημα της άμυνας. Δεν είμαι υπέρ του να ανοίξουμε ένα νέο τομέα για την αμυντική έρευνα. Υπάρχουν τόσες πολλές εθνικές επιπτώσεις εδώ πέρα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στα κράτη-μέλη για τα αμυντικά συστήματα και ζητήματα. Υπάρχουν τόσες πολλοί, τόσες άλλοι τομεί με ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία που νομίζω μπορούμε να μείνουμε σε αυτούς αντί να περάσουμε σε ένα νέο τομέα όπου προσωπικά θεωρώ ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών αποκλειστικά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή που εργάστηκε πολύ σκληρά με πιεστικές προθεσμίες και το προσωπικό που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά τόσο γρήγορα. Κατά την άποψή μου, εγώ θα ήθελα να έχω συνυπογράψει πολύ περισσότερες τροπολογίες αλλά λόγω της επιστροφής μου από το Στρασβούργο δεν πρόλαβα. Τέλος πάντων δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Το σημαντικό για εμένα είναι όταν ε, μιλάμε για την έκθεση Καρβάγιο ε, είχαμε φτάσει σχεδόν σε ομοφωνία και καμιά φορά κάποιες διατυπώσεις νομίζω μπορούσαν να είναι καλύτερες. για κάποιες τώρα από τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα αναφερθώ σε πέντε από αυτές, αν μου επιτρέπετε. Έξι, τελικά. Εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα η τροπολογία 27, που μιλάει για άλμα στην απλοποίηση. Ε, είναι αυτά τα άλματα στην απλοποίηση είναι κάτι το πολύ ωραίο. Αυτό το οποίο προβληματίζει λίγο. Η τροπολογία 1 μιλάει για την συγχρηματοδότηση. Εντάξει, μπορεί η περισσότερη συγχρηματοδότηση να χρειάζεται σε κάποια έργα, σε άλλα όμως όχι. Οπότε εγώ θα ήθελα η αυξημένη συγχρηματοδότηση να φύγει ή να πούμε όπου απαιτείται. Γιατί ε, δεν είναι μόνο θέμα συγχρηματοδότησης. Θέλω να είναι πάρα πολύ αργό για να μπουν οι λέξεις αυτές το όπου απαιτείται. Όσον μου αρέσει το υπόλοιπο, αλλά το να λέμε πως όλα χρειάζονται συγχρηματοδότηση, δεν ξέρω, ίσως παραπάει. Μετά, μιλάμε για αύξηση της χρηματοδότησης χωρίς να λέμε πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Ε, τώρα πρέπει να είμαστε λίγο ευαίσθητοι αυτούς τους καιρούς. Ε, εντάξει είμαι υπέρ της αύξησης των επενδύσεων στην έρευνα, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Φοβάμαι λοιπόν πως δεν μπορώ να υποστηρίξω την τροπολογία 26. Μιλάει για διπλασιασμό των κονδυλίων, χωρίς να πούμε πού θα βρούμε τα λεφτά. Ε, Αλλιώ δεν είμαστε πολύ αξιόπιστοι. Είναι μια διαπραγματευτική τακτική, το καταλαβαίνω, αλλά θα ήταν πιο αξιόπιστο Εάν λέγαμε και πού θα βρούμε τα λεφτά. Τροπολογία 9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει κάνει πολλά πράγματα. Να αυξήσουμε τη χρηματοδότησή του. Εάν λέγατε κιόλα ότι είναι από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 τα λεφτά, συμφωνώ. Αλλά να αυξήσουμε τις δαπάνες γενικώ με ανησυχεί. Τροπολογία 20 μετά μιλάει για την ε, ερευνητική υποδομή δεν ξέρω αν είναι γλωσσικό το σύντημα αλλά μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς λέγοντας πως ε, θα πάνε τα λεφτά στο χτίσιμο π.χ. ερευνητικών εργαστηρίων. Ε, δεν θεωρώ εγώ πως πρέπει να πάνε εκεί τα λεφτά αυτά. Πρέπει να εξοδευτούν στην έρευνα και όπου υπάρχει ανάγκη υποδομών ε, να χρηματοδοτηθεί από τα <coughs> διαρθρωτικά ταμεία να μην πάνε λεφτά από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 για υποδομές. Και επίσης η τροπολογία 11 ε, δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Εξαιρετική βεβαίως, αλλά ζητά τη σύσταση ενός κοινού συστήματος αξιολόγησης ε, της ε, έρευνας και της αριστείας και της επιδόσεως των πανεπιστημίων. Δεν ξέρω που, που πάει αυτό. Έχουμε ήδη peer reviews, εκεί πέρα βλέπουμε και την αριστεία στην παγκόσμια αγορά. Δεν ξέρω τώρα αν χρειάζεται κάτι εντός της Ευρώπης. Δεν ξέρω που το πάει δηλαδή εδώ πέρα. Να έχουμε μόνο ένα ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης της έρευνας. Δεν ξέρω. Θα ήθελα λοιπόν να σπάσει αυτή η διατύπωση, να το ψηφίσουμε χωριστά. Ίσως μπορούμε να το δούμε μέχρι να φτάσουμε στην Ολομέλεια. Η κυρία Ριέρα Εκτός μικροφώνου. Έλεγα λοιπόν πως θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του και την σκιώδη εισηγήτριά μας ε, και δυστυχώ όμω δεν μπορούσα να παρελθεί σήμερα στην συνεδρίασή μα ε, να κάνω κάποιε παρατηρήσει σχετικά με τι τροπολογίε που κατέθεσα. Κατανοώ ότι αποτελούν μέρος των ε, συμβαστικών προτάσεων που μας παρουσίασε ο Ντί. Είναι σίγουρο κύριε Σιγητά πως ε, συζητήσαμε επανειλημμένα το θέμα όπως και το θέμα της ε, απλούστευσης ε, και εγκρίναμε μια έκθεση πολύ σημαντική της κυρίας Καρβάλιο η οποία ήταν ε, πληρέστατη. Θεωρώ όμως ότι χρειάζεται να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε αυτό το σημείο χρησιμοποιώντας κάθε ευκαιρία που μας προσφέρει το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας έκθεσης τόσο σημαντική ως, αυτή της ανανεώσης του 7ου προγράμματος πλαισίου Όπως εξάλλου και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, συμφωνούν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο εμπίπτει στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Καταλαβαίνω ότι ο εισηγητής ε, δέχθηκε ένα σημαντικό τμήμα των τροπολογιών μας ε, τώρα. Κάτι ακόμα για τις τροπολογίες. Το ζήτημα του προσωπικού, του έρευνου προσωπικού. Ναι, θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό ανα πολίτες, αναπολίτη, ανακατοίκων και να υπάρχει τη συμμετοχή των γυναικών. Τώρα η έκθεση των εμπειρογνωμόνων τονίζει ότι πόρα απέχουμε από την επίτευξη των στόχων μας Φυσικά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε την συμμετοχή των γυναικών στο πλαίσιο του κύκλου ζωής ενός ε, προγράμματος. Κατανοώ πως και στο σημείο αυτό υπάρχει συμβαστική τροπολογία. Και τέλος να αναφερθώ στην πρόταση του εισηγητή σχετικά με την ε, εδαφικό χαρακτήρα των πολιτικών ε, καινοτομία και έρευνα ε, κρίνω ότι το ζήτημα είναι πολύ σημαντικά. Το εξετάσαμε επανειλημμένο στο παρελθόν. Ε, δεν πρέπει να παραιτηθούμε της αριστείας, αλλά με πολιτικές αποφάσει χρειάζεται να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα φύλλα προκειμένου όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να καταστούν άριστοι. Αυτά ήθελα να πω κύριε Οντή και συμφωνώ. πως ε, θα πρέπει το θέμα αυτό να καταστεί λίγο σαφέστερο στην έκθεσή σας. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχετε καταλήξει σε μια συμφωνία, και την οποία και θα διαβάσω πολύ προσεκτικά τώρα αναφορικά με τον αμυντικό τομέα και την έρευνα. Εμένα με ενδιαφέρει το ζήτημα της ασφάλειας όπως αυτό περιέχεται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά είμαι βεβαία ότι συζητώντας θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και περί αυτού του θέματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Καρβάλια. θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας, τον κύριο Οντή, για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε, δείξε ανοιχτό πνεύμα και δέχτηκε τις τροπολογίες μας. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που δέχτηκε το πακέτο απλούστευσης ο κύριος Οντί και δέχτηκε επίσης να συμπεριλάβει ένα κομμάτι των κατευθυντηρίων γραμμών του προγράμματος πλαίσιο 8 διότι έτσι δίνεται κάποια καθοδήγηση για το 8ο πρόγραμμα. Από πλευρά προπολογισμού, ε, υπάρχουν κάποιοι συναδέλφοι που υπέβαλαν τροπολογίε σχετικά με το dumping. Ε, ο στόχο μας δεν είναι αύξηση των δαπανών όμω. Λέμε απλώς ότι η έρευνα, κατά τη γνώμη μα είναι πιο σημαντική από άλλες πολιτικές και ζητούμε αύξηση ως εκ τούτου της γραμμής του προϋπολογισμού για την έρευνα στον επόμενο προϋπολογισμό. Ε, μία παρεμφερή τροπολογία καταθέσαμε επίσης για τον ε, γενικότερο, για το σύνολο του προϋπολογισμού. Αυτό που μένει να δούμε είναι ε, ποια, πού θα μειώσουμε τα κονδύλια, σε ποιο τομέα της πολιτικής της Ένωσης, ούτως ώστε να αντιληθούν νέα κονδύλια για την έρευνα. Αντιλαμβάνομαι ότι άλλοι συνάδελφοι ζητούν το αντίθετο. Απλώς, ξαναλέω, τονίζουμε στις ε, τροπολογίες μας ότι η έρευνα για μας είναι πάρα πολύ σημαντική για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε αυτή την τροπολογία και χαίρομαι που ε, συμπεριέλαβε την ε, τροπολογία μας αυτή στις ε, συμβαστικές του τροπολογίες, ο εισηγητής. Ευχαριστώ και θα δώσω και πάλι τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Οντί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και κυρίως τους κοιόδης εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα εντάχει να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ο κ. Τσοκαλάς δίκιο έχει κάθε φορά ευστά την προσοχή μας ε, στην, ε, στη σημασία της εκπαίδευσης και των επιστημονικών γνώσεων. Προφανέστατα είναι σημαντικό να έχουμε μια ενιαία επιστημονική κουλτούρα σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Μίλησαν κάποιοι για εδαφικότητα. Μάλλον έχω, είναι λανθασμένη διατύπωση στο, στο σημείο του κειμένου. Ο στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τους εγκεφάλους, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε όπου θα έρθουν τα νέα Νομπέλ. Οπότε σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης ε, θα πρέπει να ερευνούμε ώστε να εντοπίζουμε τους εγκεφάλους. Τώρα αναμένεται γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάμειξης από ό,τι κατάλαβα. Ε, κοιτάξτε, δεν έχω προφανώς λάβει αυτήν την έκθεση, βασίστηκα όμως σε μια ε, μελέτη για την περιφερειακή πολιτική της Επιτροπής των Περιφερειών ε, που προωθούσε αυτή την εδαφική διάσταση για την ε, πολιτική έρευνα τη Ένωση. και έχουμε την περιγραφή της συμβαστικής τροπολογίας. Ναι, μεν πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην αριστεία, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να διασυνδεθούν οι υποδομές που υπάρχουν ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς να καλλιεργήσουμε αυτή την αριστεία γιατί ε, αυτό το επιστημονικό πνεύμα είναι η προϋπόθεση εκ των όνων Ουκάνευ για να ε, δώσουμε απάντηση στις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το πρόγραμμα πλαίσιο συνδέεται έτσι και με τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα διαρθρωτικά ταμεία, ξέρετε, αποτελούν αντικείμενο μεικτής διαχείρισης με τα κράτη-μέλη. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ματίας για την υποστήριξη που μου προσέφερε. Σας ευχαριστώ για το ανοιχτό σας πνεύμα που φαίνεται από τη θέση που παίρνετε για την, στον τομέα της άμυνας και θα επανέλθω. Ε, κυρία για τη βιομηχανία, δίκιο έχετε. Ε, δεν συμμετέχουν επαρκώς ε, οι βιομηχανίες μας και υπάρχει πρόβλημα ανακολουθίας ανάμεσα στις δράσεις των κρατών μελών των βιομηχανικών ομίλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ευθυγραμμίζονται αυτές τις τρεις συνιστώσεις για να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τα χρήματα που διατίθενται για την έρευνα. Η έρευνα είναι ένας από τους τομείς όπου ναι. ε, θα έπρεπε να επιδιώκουμε καλύτερη χρήση του δημοσίου χρήματος για να στηρίξουμε ε, την βιομηχανία μας. Ο διπλασιασμός των κονδυλίων τώρα, ε, πρόταση διαφόρων συναδέλφων. Κοιτάξτε, είναι απλό σχετικά το ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να διπλασιάσουμε ε, τα κονδύλια της γραμμής αυτής. Το θέμα είναι να δούμε με ποιο τρόπο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, το πρόγραμμα πλαίσιο, την πολιτική μας για τα διορθωτικά ταμεία, πώς μπορούμε ε, όλα αυτά τα κονδύλια με συνεπή τρόπο να τα χρησιμοποιήσουμε ούτω ώστε να εξευρωπα... Ε, εξευρωπαίσουμε ε, περαιτέρω την έρευνα γιατί είναι ε, μία από τις προϋποθέσεις για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της γυραιάς Επίρου. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα ευρύτερο του διπλασιασμού των κονδύλων που διατίθεται στην έρευνα. Ας επανέλθω στον τομέα της άμυνας. Οι εμπειρογνώμονες ε, λένε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε η Ευρώπη να χάσει ή τουλάχιστον να γίνει ε, ουραγός στον τομέα αυτό της αμυντικής βιομηχανίας ε, βασιζόμενοι λοιπόν ε, στις ε, βάσεις που μας προσφέρει η συνθήκη θα αναρωτηθούμε το εξής. Για την έρευνα που σχετίζεται με την ασφάλεια ή και για την έρευνα για στρατιωτική ή μη στρατιωτική χρήση Για την έρευνα αυτή δεν πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση θα δούμε ποια θα είναι η έκβαση της αυριανής ψηφοφορίας για όλες αυτές τις τροπολογίες. Πάντως εγώ προτείνω να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα για να διαπιστώσουμε αν είναι σε θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περάσει ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή, ούτω ώστε να καταθέσει προτάσεις ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια για όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία τοποθετούμαστε επί της αρχής εμείς στο Κοινοβούλιο. Θα συνεχιστεί ο διάλογος ή του Πρόεδρε. Αυτές ήταν οι ενθερμό αντιδράσεις μου μετά από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων μου. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά. Και εμείς σας ευχαριστούμε ο Ντί για την εργασία και την προετοιμασία και αύριο ψηφίσουμε. Άρα λύεται εδώ πέρα η συνεδρίαση για σήμερα. Σας παρακαλώ λοιπόν να εγκαταλείψετε την αίθουσα γιατί θα συνεδριάσουν τώρα οι συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ.